Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ καθίστε. Euh- Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε με το εργαστήριο που προβλέπετε για την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο που μας απασχολεί παρακαλώ καθίστε και λίγη ησυχία. Ήδη έχουμε καθυστερήσει, γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε πειθαρχημένοι. Παρακαλώ. Je vous un peu de silence. Nous allons débuter, nous avons déjà du retard. Euh, cette situation au η κατάσταση στο Καραμπάχ είναι ιδιαίτερα ε, ευαίσθητη, μας, μας έχει απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του Ιουνίου είχαμε και πολλά ε, θανατηφόρα συμβάντα, δυστυχώς. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δραστηριότητα της ομάδας του Μίνσκ που προσπαθεί να επιλύσει κάπως τη διαφορά αυτή, να εξεύρει μια ευρέως αποδεκτή λύση. Τα δεδομένα όμως δεν είναι ενθαρρυντικά. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία. Ήδη πολλές φορές είχαμε εκφράσει την ανησυχία μας σε σχέση με τα λεγόμενα των δύο μερών τις στρατιωτικές προκλήσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά που αποτελούν μεγάλο κίνδυνο αναζωπήρωσης στην περιοχή. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε καταρχήν πώς έχει η κατάσταση και πώς διανοίγονται οι προοπτικές. Δεν υποκαθιστούμε τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται, ούτε και θα πάρουμε θέση σε αυτή τη θέση, σε αυτή την κατάσταση που έχει παγώσει. Απλώς θα δούμε πού βρισκόμαστε. Θα κάνουμε μία αποτίμηση. Για το εργαστήριο αυτό έχουμε μία σειρά εμπειρογνωμόνων που θα λάβουν το λόγο Tracy German από το King's College του Λονδίνου, ο κύριος Eberhard που είναι αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών στην Πολωνία, ο κύριος Ντένις Σάμουτ που είναι ο διευθυντής του Links σε σχέση με το δίκτυο αυτό για τις σειράξεις και ο κύριος Λεφόρ, ο οποίος είναι ειδικό αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο και την κρίση της γεωργίας. Εδώ έχουμε και μία αντιπροσωπεία αζέρων και ξέρετε ότι μετά την έκβαση της ακρόασης θα, έχουμε, θα συνέλθει και η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Αζερβαϊτζάν και έχουμε και παρατηρητές. Οι βουλευτές έχουν παρακολουθήσει το θέμα αυτό και θα λάβουμε το λόγο μετά από τις παρεμβάσεις των εμπειρογνωμόνων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Θα ήθελα να μιλήσουν για 12 με 15 λεπτά το πολύ, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για συζήτηση με τους βουλευτές και δίνω το λόγο στην κυρία Τζέρμαν. Thank Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την κατάσταση ασφάλειας στον Αγκόρνο Καραμπάχ και την σύραξη, η οποία δεν έχει ε, ε, επιληφθεί σε σχέση με το Αζερβαϊτζάν και την αρμενική μειονότητα, τον αρμενικό αυτό θύλακα. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες σε σχέση με το ιστορικό ή το πολιτικό σκέλος, αρκεί να πω ότι υπήρξε μεγάλη ε, διαμάχη σε σχέση με την απόφαση του Στάλιν του 20, σε σχέση με τους Αζέρους και το, τη δημιουργία αυτού, του, αυτής της δημοκρατίας Κατά το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε η σύραξη και είχαμε έναν πόλεμο ευρείας κλίμακας μεταξύ 92 και 94 με χιλιάδες θύματα και βλέπουμε, είδαμε, ότι έχουμε να κάνουμε μεγάλα τμήματα τα οποία βρίσκονται εκτός ε, του ελέγχου του Αζερμπαϊτζάν. Υπάρχει δυστυχώς, ε, δεν θα μπορούσα να πω σταθερότητα, αλλά διέξοδο και νομίζω ότι ίσως έχουν λήξει οι σειράξεις, αλλά πολλά θέματα δεν έχουν επιληθεί και υπάρχει ο κίνδυνος νέας σύραξης. Ελπίζουμε στο εγγύς μέλλον να μην έχουμε έναν ε, πόλεμο ευρείας κλίμακας, αλλά πρόκειται περισσότερο για ε, πόλεμο ελευθέρων σκοπευτών, ο οποίος όμως μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου ένας θεωρητικός των διεθνών σχέσεων μίλησε για την ε, σωστή αντίληψη λανθασμένη του ζήτηματος. Από το 2009 είχαμε μια κλιμάκωση γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ με ανταλλαγή πυρών και βεβαίως και πολλές απώλειες, πολλά θύματα πολλά ελέγχθησαν υπέρ ή κατά της παραβίασης ε, της εκεχηρίας που δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν γιατί είχαμε μόνο έξι παρατηρητές και χιλιάδες ένοπλους, άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αντικειμενική άποψη. Νομίζω ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η ανταλλαγή πυρών γινόταν σε περιορισμένους φύλακες που όλο ένα και έχουν διευρυνθεί. Αυτό το μήνα είδαμε πολλούς Αρμένιους που σκοτώθηκαν από τους Αζέρους και αυτό έγινε 30 μίλια προς βορρά της γραμμής Εκεχηρίας, δηλαδή μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Τότε ε, επισκέφθηκε την περιοχή η Χίλαρη Κλίντον η κλιμάκωση της βίας συνοδεύτηκε με αύξηση των δαπανών άμυνας και από το Αζερβαϊτζάν και από την Αρμενία και πολλά ελέγχθησαν για την κλιμάκωση απόκτησης όπλων και οι δύο χώρες δαπανούν μεγάλο μέρος του ΑΕΠ στις δαπάνες άμυνας και όλο και αυξάνονται αυτές οι δαπάνες. Το Αρμενικό Κοινοβούλιο αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 6% σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό για την άμυνα. Ως προς τις ένοπλες δυνάμεις έχω ε, έναν πίνακα στατιστικών δεδομένων. Βλέπετε ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει διπλάσιες δυνάμεις από αυτές της Αρμενίας, αλλά η Αρμενία έχει στενή σχέση με τη Ρωσία. Θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες ως προς τη... αυτούς τους συνδέσμους και εξωτερικούς παράγοντες. Η Ρωσία είναι ο πιο εύρωστος σύμμαχος της Αρμενίας που έχει στενές σχέσεις με τη Μόσχα που θεωρεί ότι βρίσκεται σε πολύ πιο ευάλωτη θέση. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Τουρκία και ένα Αζερβαϊτζάν ένα ε, και γνωρίζει μεγαλύτερη δύναμη. Ως προς τον στρατιωτικό εξοπλισμό ε, της ε, Αρμενίας, ο εξοπλισμός αυτός προέρχεται από τη Ρωσία. Υπάρχει στρατηγική εταιρική σχέση η οποία οποία ανανεώθηκε το 2010 και η ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Αρμενία απαρτίζεται, αποτελείται από 3.000 ενόπλους. Και θεωρείται ότι αυτή η συνιστός είναι πολύ σημαντική μέσα στα πλαίσια των αμυντικών δαπανών. Η Αρμενία έχει καλές σχέσεις με το Ιράν γιατί πρόκειται για μία οδό διαμετακόμισης που βρίσκεται και κοντά στα σύνορα. Πολλές ανησυχίες αναφέρθηκαν επειδή η Αρμενία συμμετέχει στη Συμφωνία Συλλογικής Ασφάλειας θεωρείται ότι η Ρωσία και άλλοι εταίροι θα μπορούσαν να προσέλθουν στην σύραξη αυτή, αλλά έγιναν πολλές δηλώσεις πρόσφατα και φαίνεται ότι αυτό δεν επίκειται. Εάν γινόταν επίθεση, δεν θα ήταν μόνο κατά της Αρμενίας και της αρμενικής περιοχής. Από πλευράς εταιρικών σχέσεων Αζερβαϊτζάν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ στενές σχέσεις με την Τουρκία που βασίζονται σε γλωσσικές και εθνοτικές ομοιότητες. Εκεί βασίζεται αυτή η συνάφεια. Υπήρχαν οικονομικές και στρατιωτικές ε, η οικονομική και στρατιωτική συμμετοχή της Τουρκίας και το 2010 το Αζερβαϊτζάν ε, συνήψε μια συμφωνία αμοιβαίας αρρωγής με την Τουρκία με στρατιωτικό εξοπλισμό σε περίπτωση επίθεσης καθώς και, ε, και συμφωνία ως προς ε, έξοδα επιμελητίας και ούτω καθεξής. Επίσης, υπάρχει ένα συμβούλιο, βαθμό συμβούλιο στρατιωτικής συνεργασίας για να προωθηθεί αυτή η συνεργασία αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Σε επίπεδο λοιπόν στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ ε, ε, Αρμενίας, Ρωσίας και Αζερβαϊτζάν, Τουρκίας βλέπουμε ότι ενισχύθηκαν αυτές οι χώρες και υπάρχει βεβαίως και ε, αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Άρα έχουμε σοβαρά προσκόμματα για την επίλυση της διαφοράς. Η Ρωσία επανέλαβε τον προηγούμενο μήνα ότι βασίζεται στις τρεις αρχές, ε, δηλαδή ε, ε, εδαφική ακαιρεότητα, αυτοδιάθεση και μη χρήση βίας, για να υπάρχει μια σχετική ισορροπία. Μας ενδιαφέρει επίσης και η πιθανότητα μεταφοράς της σύραξης στη, με βάση την γεωπολιτική σημασία των δύο χωρών και υπάρχουν και οικονομικές επιπλοκές γιατί πρόκειται για μία ε, οδό διαμετακόμισης για, προς την Κασπία ως προς τον, ε, τους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο. Και πιστεύουμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε και τις εξελίξεις στη Γεωργία, γιατί το Brent το 2008 αυξήθηκε κατά 1,5 δολάριο και τα γεγονότα του Αυγούστου 2008 στήχησαν ένα δις δολάρια σε οικονομικούς πόρους για τη γεωργία, αν και αυτό δεν λαμβάνει υπόψη και την έλλειψη εμπιστοσύνης. Μιλά μόνο για τις οικονομικές απώλειες. Άρα, η οποιαδήποτε αναζωπήρωση της διαφοράς αυτής, της σύραξης, θα είχε σοβαρές επιπλοκές. Τώρα, ως προς τους αγωγούς ε, φυσικού αερίου, υπάρχει σχετική δυνατότητα αντοχής των μέσων, αλλά ε, ελοχεύει και κάποιος κίνδυνος η κατάσταση είναι ευάλωτη και θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποια ε, σύραξη η οποία δεν είναι προβλεπόμενη, είναι τυχαία, είναι παρεμπίπτουσα. Γιατί έχουμε και μικρές αψιμαχίες, όπως γνωρίζετε, σε επίπεδο ελευθέρων σκοπευτών. Και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να προωθηθεί μία επίλυση της διαφοράς έτσι ώστε να έχουμε μία μακροχρόνια ειρήνευση της περιοχής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έμπορα έχει το λόγο. Ο κύριος Έμπορα, συγγνώμη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το τόσο επίκαιρο εργαστήριο και το λέω επίκαιρο και λυπάμαι γι' αυτό διότι η παρουσίαση δική μου θα είναι απεσιόδοξη θα έλεγε. Καταρχάς ε, παρουσιά, βλέπουμε ότι υπάρχουν εντάσεις, ιδίως ε, υπάρχει μια τεταμένη ατμόσφαιρα και όσον αφορά την ε, κατάπαυση του πυρός και υπάρχουν προβλήματα και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο κοινής γνώμης και στο Αζερβαϊτζάν και στην Αρμενία. Δεύτερον, ε, στο δεύτερο κομμάτι ε, ε, είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να επιληθεί το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχα. Και εάν παραμείνει η κατάσταση ως έχει, σε κάποια χρόνια θα ξαναρχίσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και έναν τυχαίο πόλεμο στην περιοχή. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή όμως. Ε, ενδιαφέρει το Καραμπάχ. Έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχει οικονομικούς πόρους, δεν έχει φυσικούς πόρους, δεν έχει στρατηγική σημασία. Μεν. Όμως έχει συμβολική και ιστορική σημασία και για το Αζερμπατζάν και για την ε, Αρμενία. Είναι το λίκνο, το βασικό λίκνο και για το Αζερβαϊτζάν και για την Αρμενία. Και όλη αυτή η, η συμπλοκή και οι εχθροπραξίες που παραμένουν, που παραμένει, ε, επηρεάζει τις ζωές και των δύο χωρών. Ας δούμε το Αζερβαϊτζάν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Αζερβαϊτζάν έχει χάσει κατά διάρκεια του πολέμου το 16% της επικράτειάς του. Και αυτό εμφανίζεται σαν μια εμφανής αδυναμία του κράτους. Η διαμάχη στο Καραμπάχα έχει δημιουργηθεί σαν, και χρησιμοποιείται μάλλον από την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν σαν ένα στοιχείο ε, ένωσης ε, του κράτους και εμφανίζεται και η μεγάλη σφαγή του 1992 σαν η στη σφαγή του Χοτζάλι Μαχάλ βλέπετε εδώ στην διαφάνεια, σε ένα, σε ένα δρόμο του Μπακού που έγινε η μεγάλη ε, εκδήλωση μνήμης ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι οι πρόσφυγες. Έχουν ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων από το Καραμπάχα. Είναι το 8% του πληθυσμού του Αζερβαϊτζάν. Δεν έχουν ενσωματωθεί όμως στην κοινωνία και αυτή η απομόνωση των προσφύγων είναι η εσωτερική πολιτική, οφείλεται η εσωτερική πολιτική της κυβέρνησης, διότι τους ε, ε, συμφέρει να υπάρχει αυτός ο αριθμός των προσφύγων για να πιέσουν τη διεθνή κοινότητα, για να δείξουν ότι εάν δεν επιληθεί και όσο δεν επιλύεται η διαμάχη του Ναγκόρνο Καραμπάχ υπάρχουν προβλήματα. Τώρα ζούμε την, ε, την κατάσταση από την πλευρά της Αρμενίας θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτός ο νικητήριος πόλεμος, η νίκη τους δηλαδή στον πόλεμο του Καραμπάχα, είναι ένα στοιχείο εθνικής υπερηφάνειας και είναι από τα κάποια στοιχεία αν θέλετε ε, εθνικής υπερηφάνειας και σύγχρονης ταυτότητας και είναι ένας παράγοντας ε, κοινωνικής ε, ολοκλήρωσης. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι η επίλυση της διαμάχης στον Ακόρνο Καραμπάχα για το... είναι πολύ πιο σημαντική για την Αρμενία. Η Αρμενία είναι ανάμεσα στην Τουρκία, βρίσκεται ανάμεσα στην Τουρκία και στο Αζερβαϊτζάν και είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να διατηρήσουν υποέλεγχο τον Ακόρνο Καραμπάχα και όχι να βρουν μια συμβαστική λύση με τους γείτονές τους. Και τα τελευταία 20 χρόνια η Αρμενία βρίσκεται σε μια περιφερειακή ή μη απομόνωση θα τη χαρακτήριζα. Βλέπετε μια εικόνα, βλέπετε Είναι, είναι, αυτή είναι μια φωτογραφία από μια στάση του λεωφορείου και είναι ο χάρτης της Αρμενίας και φαίνεται και τον Ακόρνο Καραμπάχα, είναι κοινή φωτογραφία αυτή και βλέπετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει τον Ακόρνο Καραμπάχ στην Αρμενία αλλά η εικόνα δεν είναι και τόσο σαφής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στην Αρμενία και στο Καραμπάχα. διότι η Αρμενία τουλάχιστον δεν έχει αναγνωρίσει την, ανεξαρτησία του Καραμπάχα. Ταυτόχρονα όμως η Αρμενία εκπροσωπεί το Καραμπάχα στην ειρηνευτική διαδικασία. Ε, εφόσον το Αζερβαϊτζάν εμποδίζει τον Ακόρνο Καραμπάχ να συμμετέχει στο τραπέζι των ε, ε, διαπραγματεύσεων. Ε, η, η Αρμενία υποστηρίζει πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά το Καραμπάχ. Υπάρχουν κοινωνικοί δεσμοί, αλλά ταυτόχρονα παρά την ανεξαρτησία την, και την ε, εξάρτηση ε, ανάμεσα στην Αρμενία και στο Καραμπάχ, δεν μπορούμε να πούμε ότι η, ότι η κυβέρνηση του Καραμπάχα πρέπει να σέβεται όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ερεβάν. Η Αρμενία ε, η Αρμενία κληρονόμησε όλη την ελίτ την κυβερνητική από το Καραμπάχα. Και ο πρόεδρος της Αρμενίας ήταν παρόν σε μια στρατιωτική παρέλαση στον Ακόρνο Καραμπάχ πριν από ένα μήνα για να γιορτάσουν το τέλος του πολέμου, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, αλλά και την ε, ε, κατάληψη πριν από 20 χρόνια μιας ε, πόλης της πόλης Σουσία από τις αρμενικές δυνάμεις στον Ακόρνο Καραμπάχ. Τώρα ας δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ποιε είναι οι θέσεις των κρατών. Το Αζερβαϊτζάν τι λέει ότι θα πρέπει να επανέλθει ο έλεγχος για τις αμφισβητούμενες περιοχές και ότι ο, ε, ο, λαός, οι πολίτες περιμένουν ότι θα ξαναρχίσει ο πόλεμος με την τελική νίκη του Αζερβαϊτζάν. Η Αρμενία θεωρεί ότι ε, η, η διαμάχη αυτή, ο πόλεμος αυτός έχει ήδη ε, τελειώσει και δεν, δεν έχουν καμία πρόθεση να ζητήσουν μια κάποια συμβαστική λύση με το Αζερβαϊτζάν. Επίσης, η, Επίσης η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ούτε θέλει ούτε μπορεί όμως και να αγνοήσει την κοινή γνώμη. Ενώ η αντίστοιχη κοινή γνώμη της Αρμενίας ε, δεν ε, θέλει, δεν, έχει, δεν θεωρεί ότι υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις. Επίσης το πρόβλημα είναι ότι ε, ένα μεγάλο ποσοστό των Αρμενίων που διαμορφώνουν και την κοινή γνώμη, ζει εκτός της Αρμενίας. Άρα δεν ε, υφίσατε τις συνέπειες της ημιαπομόνωσης της χώρας. Τώρα, η ισορροπία των δυνάμεων. Το, ε, το έχει έσοδα από τα πετρέλαια. 20 δισεκατομμύρια το 2011 και αυξάνεται στρατηγικό, η στρατηγική σημασία της χώρας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία και την Ρωσία. Επίσης, οι στρατιωτικές δαπάνες 3 δισεκατομμύρια το 2011 σε σχέση με τα 130 εκατομμύρια το 2003. Οι στρατιωτικές δαπάνες ε, για το Αζερμπαϊτζάν το 2012 θα είναι 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια είναι δύσκολα να τα συνειδητοποιήσει κανείς αυτά τα ποσά, διότι οι στρατιωτικές δυνάμεις κατανέμονται στις ε, διάφορες, ε, στα διάφορα κυβερνητικά κονδύλια, στα διάφορα κονδύλια δημοσίων δαπανών. Παρόλα αυτά όμως οι στρατιωτικές δαπάνες στο Αζερβαϊτζάν είναι, είναι μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό, το συνολικό προϋπολογισμό του ε, της Αρμενίας και είναι 8 ε, φορές παραπάνω από τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της Αρμενίας και του Καραμπάχ ε, μαζί. Ένας μεγάλος προμηθευτής όπλων του Αζερμπαϊτζάν είναι το Ισραήλ. 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια συγγνώμη, είναι το τελευταίο συμβόλαιο που υπογράφηκε και βλέπετε ότι Υπάρχει ε, ψωμί εδώ αν θέλετε. Το Αζερμπαϊτζάν έκανε την ε, μεγαλύτερη πραγματική ε, ποσοστία αύξηση στις στρατιωτικές δαπάνες ε, σε όλο τον κόσμο 2011. Όπως λέει το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης. Το Αζερμπαϊτζάν τώρα αισθάνεται ότι η εξουσία του, η δύναμή του δεν συνοδεύεται από κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις στο Καραμπάχ. Και ο πολιτικός κόσμος ε, και αισθάνεται μία απογοήτευση. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και μία μιλιταριστική προπαγάνδα και η κοινή γνώμη αισθάνεται κουρασμένη. Και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση γίνεται όμοιρος της κοινή ε, γνώμης. Κοινή γνώμη την οποία η ίδια έχει διαμορφώσει. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι στην Αρμενία υπάρχει και ένα κλίμα επιβίωσης αν θέλετε Έχουμε περισσότερες ε, εντάσεις και δεν θέλουν ούτε οι Αρμένοι ούτε οι Αζέροι να, να κάνουν οποιαδήποτε παραχώρηση. Σας είπα για την ε, δύναμη της, ε, της συνέστηση εξουσίας και δύναμης που έχει το Αζερβαϊτζάν. Αναφερόμαστε και τώρα και σε μία δήλωση του Προέδρου Αλίεγεφ, ο οποίος λέει ότι η η υπομονή μας ε, εξαντλείται, δεν είναι ανεξάντλητη και ότι αν δεν ε, αποδώσουν ε, οι διαπραγματεύσεις τότε θα ξαναρχίσει ο πόλεμος και θα είμαστε τότε έτοιμοι. Αυτά τα είχε πει το 2007 αλλά τέλος πάντων και τώρα στα ίδια πράγματα πιστεύουν. Τώρα, Τελευταία ερώτηση που έκανε ο πρόεδρος Αλίεγεφ. Λέει, είναι έτοιμο το Αζερμπαϊτζάν. Όμως, είναι. Καταρχάς, οι Αρμένοι είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην ε, σύγκρουση αυτή στον Καραμπάχα, διότι ελέγχουν τις αμφισβητούμενες περιοχές, έχουν ισχυρή στρατιωτική δύναμη και έχουν την πολιτική και ε, στρατιωτική υποστήριξη από την Ρωσία. Τώρα, αν πάρουν όμως οι Αζέρι τα όπλα από το Ισραήλ, το πρόβλημα θα, είναι, θα τεθεί με διαφορετικούς όρους. Αν δούμε τώρα και την θέση της Αρμενίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο τις στρατιωτικές δυνάμεις της, αλλά και την υποστήριξη της Ρωσίας το Καραμπάχ είναι το πιο ισχυρό όπλο και εργαλείο που διαθέτει η Μόσχα στην πολιτική ε, απέναντι στο Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Υπάρχει μια εμπλοκή του πρώην Προέδρου Μετβέντεφ για την επίλυση του προβλήματος. Τελικά όμως δεν κατάφερε να πετύχει ο Πρόεδρος. Πιστεύουμε ότι η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί η μονομερή επίλυση του προβλήματος. Ταυτόχρονα όμως μία ενίσχυση των ε, εντάσεων μπορεί να ευνοήσει και τη Ρωσία κιόλας. Υπάρχει και ένα δύναμο σημείο για το Αζερμπαϊτζάν ποια, η δύναμη που έχει το Αζερβαϊτζάν στηρίζεται απόλυτα με την δυνατότητα εξαγωγής του πετρελαίου της. Εάν βομβαρδιστεί ένας αγωγός, εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, έχουν, υπάρχουν πολλοί ο, αγωγοί που ξεκινούν από τον Πακού, πηγαίνουν στην Τυφλίδα, στο Νοβοροσυρίσκ. Ε, αν γίνει οτιδήποτε εκεί, τότε καταραίει το όλο οικοδόμημα. Λοιπόν, να συνοψίσω. Έχουμε αυξανόμενες εντάσεις. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ε, τα πρόθυρα ενός πολέμου αλλά και αυτό να μην ε, σημαίνει ή ασκούνται πιέσεις στην Αρμενία και την διεθνή κοινότητα να παραμείνει το Καραμπάχ στην ε, διεθνή ατζέντα. Και πιστεύουμε ότι ο πόλεμος είναι μια ε, εναλλακτική λύση που αποτελεί κίνδυνο για την πολιτική ελίτ του Αζερβαϊτζάν, διότι καταρχάς μάλλον δεν θα εξασφαλίσει την φιλική ουδετερότητα της Ρωσίας στον Πακού και μία ήττα θα δημιουργήσει και ένα κίνδυνο για μία διεθνή ε, κατάρρευση. Τώρα, ποιες είναι οι προοπτικές. Καταρχάς, ε, φαίνεται ότι το Αζερμπαϊτζάν μπορεί να ξεκινήσει ένα πόλεμο μεγάλης, ε, μεγάλης κλίμακας. Θα ήθελε όμως το πρόβλημα είναι ότι μία στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα εφόσον υπάρξει μια αλλαγή στην ισορροπία των δυνάμεων και ένας τυχαίος πόλεμος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Έστω δηλαδή και αν η δέσμευση της διεθνούς κοινότητας σήμερα είναι να μην γίνει πόλεμος ε, και πρέπει αυτή την άποψη η διεθνής κοινότητα να την επιβάλλει αν δεν θέλουμε να ξεσπάσει ένας πόλεμος αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής. Ο κύριος ε, Σαμί. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ κυρίως ε, στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν ε, την σύγκρουση. Θα ήθελα να πω και μερικά πράγματα για το πλαίσιο Καταρχάς, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι παρόλο που το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχα υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 25, 25 ε, χρόνια, ε, η φύση του έχει αλλάξει. Άρχισε ως ε, εθνοτική διαμάχη στα τέλη του 1980 και τώρα έχει φτάσει να είναι μια σύγκρουση μεταξύ δύο ανεξαρτήτων κρατών, της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν. Η, περιφέρεια, η περιοχή αυτή, όπως είπαμε, είναι μεγάλη στρατηγική σημασία ε, ε, ε, στις ενεργειακές οδούς από την Κεντρική Ασία και την Ευρώπη, συνορεύει με την Ρωσία, την Τουρκία και επομένως πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν σημαντικές οικονομικές, θρησκευτικές και πολιτικές σχέσεις με την περιοχή. Το βασικό πρόβλημα τώρα είναι το θέμα της ασφάλειας, η ασφάλεια του πληθυσμού, της της ε, περιοχής. Ε, κάθε επίλυση ε, του προβλήματος πρέπει να λάβει υπόψη την ασφάλεια της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, όπως επίσης και, των, και εξωτερικών μερών αν μία ακόμη φορά υπάρξει σύγκρουση θα είναι πολύ πιο θανατηφόρα από ότι ε, στις αρχές της δεκαετίας του 90 και όπως αναφέρθηκε ε, ε, υπάρχουν όπλα στην περιοχή και η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση ετοιμότητας σήμερα για πόλεμο από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν ότι ο κίνδυνος κλιμάκωσης κρίσης είναι πλέον υψηλό, είναι μεγάλος ε, είναι πλέον μια γειτονική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας ενδεχόμενος πόλεμος θα πλήξει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την ανάγκη ε, να παραμείνει ανοιχτή η περιοχή ως πύλη ε, για ε, τις ενεργειακές οδούς. Αυτό μπορεί να έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση που θα προκύψει. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος αν τρίτα μέρη ε, συμμετέχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην όλη σύγκρουση. Επομένως είναι προ συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λυθεί το συντομότερο δυνατόν το πρόβλημα φαίνεται όλο και περισσότερο ότι δεν είναι ικανοποιητικό απλώς να γίνεται ανάσχεση της σύγκρουσης ε, γιατί δεν είναι παγωμένη αυτή η σύγκρουση. Πεθαίνουν ε, στη γραμμή ε, των συνόρων όλο και περισσότεροι και η κατάσταση είναι πλέον μη βιώσιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να εμπλακεί σε σημαντικές προσπάθειες για μια μακροχρόνια λύση, κάτι το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντικα να αντικαταστήσει τους μηχανισμούς ε, του 1992 για ε, διαμεσολάβηση στην, κρίση. Ε, όμως σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει όρους για την υποστήριξή της. Μετά από 20 χρόνια είναι σημαντικό να αναμένει κανείς μία αναθεώρηση της, των μηχανισμών. Μπορεί όμως η Ένωση να βοηθήσει την ελληνευτική διαδικασία χωρίς να είναι ένας άμεσος παίκτη Υπάρχουν κάποια μέσα αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ε, γραφείο του ειδικού ε, απεσταλμένου με τη βοήθειά του μάλιστα δύο σημαντικά πράγματα συνέβησαν. Πρώτον, ε, είναι πολύ σαφέστερη η εντολή ε, όσον αφορά ε, την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότιο Κάφκασο και στις σχετικές συγκρούσεις όπως αυτή του Ναγκόρνου Καραμπάχ και επίσης ο ειδικός απεσταλμένος έχει ιδιαίτερη πείρα για την στην περιοχή, κάτι το οποίο είναι πολύ ε, σημαντικό όταν τίθεται στο επίκεντρο των πραγμάτων. Και το ε, Κοινοβούλιο ε, έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί και με τις δύο πλευρές και έχουμε δει ότι υπήρξαν σημαντικές συνεδριάσεις και στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν. Θεωρώ ότι ήταν σημαντικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και επίσης μετά από πολλά χρόνια αναμονής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιπροσωπείες που εργάζονται και στις δύο περιοχές και ε, συμμετέχει ενεργά και στις διαπραγματεύσεις και με τις δύο πλευρές. Υπάρχουν επίσης μηχανισμοί κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της ανατολικής ε, ε, συνεργασίας κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει την επίλυση του προβλήματος. Νομίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στην ισχύ διαφόρων στοιχείων ε, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι ε, προσπάθειες ε, είναι συμπληρωματικές. Θα ήθελα να μιλήσω και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης γιατί ακούσαμε πολλά για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη των μέτρων αυτών ως συνεισφορά στην ειρηνευτική διαδικασία. Αυτό είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη βεβαίως, όμως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και πολύ καλά τι σημαίνουν αυτά τα μέτρα, τι είναι και τι μπορούν να επιτύχουν και τι δεν μπορούν να επιτύχουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ε, είτε για τους πολίτες είτε στρατιωτικά, ε, δεν πρέπει να είναι υποκατάστατο μιας ε, αξιόπιστης ειρηνευτικής διαδικασίας, πρέπει να συμπορεύονται με την ειρηνευτική διαδικασία αυτή καθεαυτή. Και όπως κατέστησε αφές από τον Υπουργό Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν την περασμένη εβδομάδα, μία από τις δύο πλευρές δεν είναι έτοιμη να δεχθεί αυτά τα μέτρα, εάν τα θεωρούν τμήμα ε, παγίωσης ε, της τρέχουσας κατάστασης, παρούσας κατάστασης, του status quo. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό αυτά τα μέτρα να δίνουν τη δυνατότητα και στις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν. Το πώς μπορούν να εφαρμοστούν ε, δεν ε, έχει όριο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προβεί σε τέτοιου είδου μέτρα, πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα και στι δύο πλευρέ που θα. Ε, ε, ε, μια, μια κατάσταση που θα μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα διαπαντό. Είναι πολύ σημαντικό τα μέτρα αυτά να ε, μην δίνουν περιθώρια παρανόησης, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες ε, συνθήκε για τις διαπραγματεύσεις, ώστε αυτές να είναι επιτυχείς. Αν λοιπόν φτάσουμε στις διαπραγματεύσεις, τότε τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποκρισταλώσουν μια ε, συμφωνία, όμως σε κάθε περίπτωση τα μέτρα οικοδόμηνης εμπιστοσύνης πρέπει να εξετάσουν τις διάφορες πτυχές του προβλήματος και σε επιτόπου επίπεδο και με τις πληγήσεις ε, ε, περιοχές ε, όπως επίσης και να μην εκφυλιστεί ο διάλογος στις δύο κοινωνίες για το θέμα αυτό. Πρέπει να δούμε επίσης και την ασφάλεια των, των θα ήθελα να πω ότι έχω 10 συστάσεις ε, δράσεων που μπορούν να αναλυφθούν ε, για την επίλυση του προβλήματος από τον εσωτερικό συντονισμό των ε, προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετοχή στρατιωτικής φύσεως, κάλυψη του επικοινωνιακού χάσματος, όπως επίσης και μια πραγματική προσπάθεια περιφερειακής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται για πολλά από αυτά να περιμένει κανέναν, μπορεί να δράσει μονομερός. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλό να υπάρχει συγκατάθεση και των δύο πλευρών. Κύριε Πρόεδρε, εδώ τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται προβληματικά παρά το γεγονός ότι υπήρξαν γενικές δηλώσεις εκτίμησης ε, της ε, υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση του προβλήματος του Καραμπάχ, ε, πρέπει να είναι πολύ σαφέστερα τα μηνύματα από τις κυβερνήσεις Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν ότι θέλουν μια συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση της διαμάχης και κυρίως για τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Πρέπει να τα ακούσουμε αυτό καθαρότατα. Υπάρχουν κι άλλοι, θα μπορούσαμε να πούμε, ε, εκτός από τις δύο πλευρές της διαμάχης, που δεν ε, συμφωνούν ιδιαίτερα με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είναι λοιπόν σαφές ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την επίλυση του προβλήματος, ειδικότερα αν και η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν το επιθυμούν. Κύριε Πρόεδρε, η διαμάχη αυτή στον Αγκόρνο Καραμπάχ δημιουργεί ένα πρόβλημα ε, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες, ε, αντίκτυπο πολύ πέρα από την περιοχή. Ένα ανεπίλητο, μια ανεπίλητη σύγκρουση ε, υπονομεύει στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό χρειάζεται στεναρή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λυθεί το πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά του, χωρίς να συμμετέχει υποχρεωτικά στην ειρηνευτική διαδικασία και στον ε, μηχανισμό διευκόλυνσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Μετά από όλες αυτές τις ε, διαπιστώσεις, ε, μάλλον αρνητικής φύσεως, υπήρξαν βέβαια κάποιες δίωδη επίλυση του προβλήματος, να δώσουμε και το λόγο στον Φιλίπ Λεφόχ, που είναι ο ειδικό απεσταλμένος Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μας πει ορισμένα πράγματα για το τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε, να, να ανταποκριθώ χρησιμοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα εχμής που διαθέτουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Euh, Τρία σημεία θα ήθελα να θίξω. Καταρχήν, ορισμένα βασικά στοιχεία ως προς την ειρηνευτική διαδικασία που θα πρέπει να υπενθυμίζουμε από καιρού εις καιρών. Για να ξέρουμε ε, ακριβώς γιατί μιλάμε. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να υπενθυμίσω αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η δική μας αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και της ενδεχόμενες εξελίξεις. Η ειρηνευτική διαδικασία έχει αναλυφθεί από την ομάδα του Μίνσκ και δεν έχει συνέλθει ποτέ στο Μίνσκ. Πρόκειται για έντε χώρες που απορτίζουν την, στις χώρες της ειρήνευσης που δεν συνήλθαν ποτέ στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Το 1992-1994 είχαμε μία ευρύτατη σύραξη και στη συνέχεια ανακοχή που διαπραγματεύτηκε η Ρωσία Μετά από το 1996 είχαμε μία συμπροεδρία που ορίστηκε και που περιελάμβανε τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία και την Ρωσία και την Ομοσπονδία της Ρωσίας. Πρόκειται για μια πολιτική συνεργασία γιατί βλέπουμε ότι οι αρχηγοί κρατών ασχολούνται με το θέμα μέσα στα πλαίσια της Συνπροεδρίας. Σε πρώτη φάση οι Αμερικανοί το 98-99 όπου σχεδόν καταλήξαμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Στη συνέχεια όμως δολοφονήθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας στην Αρμενία, κάτι το οποίο δείχνει ότι οι επικεφαλής κρατών αναλαμβάνουν κινδύνους. Στη συνέχεια είχαμε τη γαλλική φάση υπό τον ε, Σιράκ το 2002, 2003 και 2004 και από το 2010 μπαίνουμε στη ρωσική φάση όπου συμμετείχε και ο πρόεδρος Μεντβέντεφ κατά τις συνεδριάσεις του 10-11 μέχρι και τις αρχές του 12. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι η διαδικασία αυτή οδήγησε σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο, ένα προσχέδιο. Πρόκειται για τις αρχές της Μαδρίτης, διότι καταρτίστηκαν για πρώτη φορά στη Μαδρίτη και μετά επανασυντάχθηκε το σχέδιο και υπάρχουν, υπάρχει και ένα σκέλος συμφωνίας που είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Το περιεχόμενο εκφράστηκε δημοσίως από τους τρεις επικεφαλής κρατών το 2010 στους G8 της Άκουιλα. Πρόκειται για έξι αρχές και καλό θα ήταν να έχετε και το χάρτη μπροστά σας, δηλαδή επιστροφή των κατεχομένων του Ναγκόρνο Καραμπάχ κοντά στο σοβιετικό, το πρώην σοβιετικό μπλάστ του Άνω Καραμπάχ προς Ανατολάς. Ανατολικά του Ναγκόρνο δηλαδή. Οι Αρμένοι μιλάνε για ζώνη ασφαλείας και η ομάδα του Μίνσκ μιλάει για κατεχόμενα. Αυτή είναι η πρώτη αρχή. Η δεύτερη αφορά ένα ενδιάμεσο καθεστώς για τον Αγκόρνο Καραμπάχ μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας και της αυτοδιάθεσης και αυτοδιακυβέρνησης. Ένας δίευλος που να συνδέει την Αρμενία μεταξύ, ε, ε, που να συνέει την Αρμενία με τον Αγκόρνο Καραμπάχ, στο Άνω Καραμπάχ δηλαδή, εκεί που σας δείχνω, ήδη υπάρχει ένας δρόμος που έχει διανοιχτεί. Εδώ ορίζεται ο διάβλος, ένα τελικό καθεστώς για τον Αγκόρνο Καραμπάχ που θα οριστεί στο μέλλον με την ελεύθερη βούληση των λαών που θα είναι δεσμευτική. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει η λέξη δημοψήφισμα εδώ. Για εύλογους λόγους, ούτε γίνεται λόγος για αυτό διάθεση. Το δικαίωμα όλων των εκπατρισμένων να επανέλθουν και τις διεθνείς συνθήκες ασφαλείας, μια διεθνή συνθήκη περί ασφάλειας που να αφορά ε, έναν δίευλο ειρήνευσης και επικοινωνίας. Βέβαια, ο διάβολος βρίσκεται στο, στις λεπτομέρειες. Αυτός ο διάβολος πού θα βρίσκεται και πώς θα ορίσουμε για το μέλλον την ε, ελεύθερη έκφραση, τη λαϊκή ελεύθερη έκφραση στο εγγύς μέλλον. Τι είναι το εγγύς μέλλον, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, ποτέ ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή μεταξύ της επιστροφής των εκτοπισμένων και των προσφύγων και του ορισμού ενός ε, τελικού καθεστώτος για το Άνω Καραμπάχ. Αυτά όλα συζητήθηκαν στα πλαίσια της ομάδας του Μίνσκ, εντός και εκτός, και εδώ βρίσκεται το όλο διακύβευμα της διαπραγμάτευσης. Τώρα, ως προσθέσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην όλη διαδικασία. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται. Πρόκειται για δύο βασικά κείμενα που αποτελούν τον οδικό χάρτη που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Δευτέρου του 12 και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Ψήφισμα της 18ης Απριλίου 2012 και θα σχολιάσω και τα δύο κείμενα σε ένα λεπτό. Αυτό είναι ένα από τα μέσα Έχουμε και το, την ύπατη εκπρόσωπο βεβαίως και τα προγράμματα που έχουν ε, στη διάθεσή τους τα συμβαλόμενα μέρη, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επίσης το ευρωπαϊκό πρότυπο βασίζεται στο συμβασμό και στην εξέβρεση πραγματιστικών λύσεων υπέρ των λαών που έχουν πληγεί από την ένοπλη σύραξη για να αλλάξει και η ατμόσφαιρα και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε πολιτικές λύσεις, ιδιαίτερα σε τομείς όπου δεν φαίνεται εύκολη η πολιτική λύση από τον ανταγωνισμό που υπάρχει. Αυτοί οι μηχανισμοί και τα μέσα θα ήταν χρήσιμα για τα εμπλεκόμενα μέρη. Έγινε λόγος για διπλά πρότυπα, δεν υπάρχουν και το τονίζω αυτό, βασιζόμαστε στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, στις αρχές του Ελσίνκη και το Χάρτη των Παρισίων, Βεβαίως οι καταστάσεις διαφέρουν μεταξύ σειράξεων στη Γεωργία, στη, στα Βαλκάνια και στο Άνω Καραμπάχ. Θα ήθελα όμως να πω σαφέστατα ότι τηρούμε τις ίδιες αρχές σε όλα τα σημεία του κόσμου. Αυτή είναι και η βασική μας γραμμή. Ως προς τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα γνωρίζετε και θα τα θυμόσαστε. Είναι επίκαιρα. Η μεγάλη μας ανησυχία για την μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν η υποστήριξη της ομάδας του Μίνσκ, και, του Μίνσκ και των αρχών της Μαδρίτης μετά, και σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα έπρεπε να δούμε κατά πόσο θα αλλάξει η σύνθεση, δηλαδή κατά πόσο θα πρέπει να αντικατασταθεί η Γαλλία. Κρίναμε και εδώ είναι συνενετικό το σχήμα μας. Συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα ότι θα πρέπει να μην ανοίξουμε αυτό το κουτί της Πανδώρας ως προς την σύνθεση της ομάδας του Μίνσκ. Δεν θα είχε νόημα να μιλάμε για τη διαδικασία, μας ενδιαφέρει η ουσία. Δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο αυτή την συνενετική διαδικασία της Μαδρίτης γιατί θα χάναμε το σωστό ορίζοντα, κάτι το οποίο δεν μας επιτρέπεται. Οι εμπειρογνώμονες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σε σχέση με τις εντάσεις που υπάρχουν στην διαχωριστική γραμμή, κάτι το οποίο συμμερίζονται και τα θεσμικά όργανα. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πρόσφατο, ε, πρόσβαση με συγχωρείτε, στο, στη συμμετοχή ως προς αυτό το συνενετικό σχήμα, χωρίς όρους. Ανεφόρον λοιπόν πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, αντιπροσώπων της. Για αυτή την ε, πρόσβαση δεν έχουμε εντολή. Ο ΑΣΕ έδωσε εντολή στην ομάδα του Μίνσκ να μπορεί να προβαίνει σε προτάσεις, να εκφράζει επιθυμίες των ε, συμπλεκομένων μερών, των εμπλεκομένων μερών για να δούμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση. Δεν έχει νόημα να μιλάει κανείς για το Άνω Καραμπάχα, αν δεν έχει μεταβεί ποτέ. Επίσης θεωρούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουμε να κάνουμε με μία ε, γενναιόδαρη πρόταση η οποία δεν την, δεν την είχαν υποστήριξης παρά από την ε, διεθνή κοινότητα γενικά. Ένα από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στο Λοσκάμπος χτες η ομάδα του Μίνσκ αναφέρθηκε για τα ευεργετήματα ενός ε, ε, Κάφκασου ειρηνικού που διαβεί υπό ειρηνικές συνθήκες για να δούμε ποια θα είναι τα ευεργετήματα, τα οποία είναι πολλά και για όλους, ανοικοδόμηση του Καυκάσου, επίσης κάτι το οποίο θα είχε μεγάλη σημασία. Μετά από τα Βαλκάνια πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία. Πρόκειται για ένα προσχέδιο ανοικοδόμησης του Καυκάσου, που θα αποτελέσει και την ε, δική μας συνεισφορά στην επίλυση της ε, διαφοράς αυτής. Ως προς τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, τα γνωρίζετε πολύ καλά, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και η ΕΕΔ, θα πρέπει να προβούν σε εύλογες συμφωνίες και διαβουλεύσεις σε σχέση με τις συμφωνίες σύνδεσης και ούτω καθεξής. Μιλάμε για την ανάγκη να υπάρχει η σωστή μόχλευση το σχέδιο το γνωρίζετε, είναι οι αρχές της Μαδρίτης και θέλουμε να ξεφύγουμε από τον πόλεμο, από την εμπόλεμη κατάσταση και θέλουμε ακριβώς γι' αυτό το λόγο να δείξουμε τα πλεονεκτήματα στους πολιτικούς και στους πολίτες. Έτσι ώστε να επιληθεί η σύραξη και από τις δύο πλευρές. Επρόκειτο για ένα σαφές μήνυμα προς τις αρμόδιες αρχές. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με τις ε, λεπτομέρειες ως προς την εντολή, ως προς την ε, τρέχουσα κατάσταση. Ε, έγινε λόγος για κίνδυνο μακροχρόνια σύραξης. Ο κίνδυνος δεν είναι άμεσος. Υπάρχουν φάσεις έντασης με θύματα ο, η βία και ο κίνδυνος βίας είναι πολύ υψηλός. Δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε μια στρατιωτικοπολιτική σύραξη υψηλής έντασης. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο διατρέχουμε κίνδυνο τυχαίου πολέμου με βάση την γεωπολιτική κατάσταση. Πρόκειται για μια ενδυνάμει ε, κατάσταση η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει την διεθνή κατάσταση τη, με βάση τις συγκεκριμένες συγκυρίες που διαγράφονται. Η κάθε χώρα και οι δύο χώρες ε, έχουν να αντιμετωπίσουν τις αρχές της Μαδρίτης που ίσως αποτελούν ένα επώδυνο σχέδιο και βλέπουμε για το Αζερβαϊτζάν ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση υπεροχής. Άρα ο χρόνος ε, τάσεται, συνδράμει τους Αζέρους περισσότερο και από πλευράς Αρμενίας υπάρχει μια αντίσταση και ένα status quo που σχετίζεται με το συλλογικό, τη συλλογική ψυχολογική κατάσταση και το συλλογικό υποσυνείδητο των Αρμενίων, στο οποίο δεν θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα. Τι μπορούμε να κάνουμε έμπρακτα να μην απελπιστούμε σε πρώτη φάση. Έχουμε να κάνουμε με μια ειρηνευτική διαδικασία, η οποία δεν είναι σαν μια, εμπορική ε, συναλλαγή. Έχει συναισθηματική φόρτιση. Υπάρχουν φάσεις ε, απελπισίας, φάσεις ελπίδας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό αφορά και την ε, δυνατότητα αποσόβησης ενός ε, μιας στρατιωτικής ε, σύγκρουσης. Διαφορετικά αρχίζουμε από το μηδέν. Η εργασία μας θα πρέπει να είναι συλλογική μαζί με τους διαμεσολαβητές της ομάδας του Μίνσκ έτσι ώστε να γνωρίζουν οι λαοί ότι υπάρχουν ε, εναλλακτικές ε, οδοί από το να σκοτώνονται και ιδιαίτερα νέοι από ελεύθερους σκοπευτές. Και υπ' αυτή την έννοια υπάρχουν δύο μέσα. Τα στρατιωτικά μέσα οικοδόμησης εμπιστοσύνης Θεωρητικά και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη θεωρούν ότι θα πρέπει να ε, ανοίξει μία έρευνα στην γραμμή επαφής και η επανάληψη ενός διαλόγου και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είναι ανύπαρκτα αυτή τη στιγμή. Τρίτον, να δείξουμε ότι τα ευεργετήματα μιας ειρήνης είναι κάτι το απτό και ιδιαίτερα θετικό και για τις δύο χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Τσαμπογνόρ θα, ήθελα να, θα θέλαμε να μας πει λίγα λόγια γιατί προεδρεύει της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και την Γεωργία. Θέλετε να πάρετε τώρα το λόγο και μετά στους υπόλοιπους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να τονίσω ότι και οι δύο χώρες είναι σημαντικές και ισότιμοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Ξέρω ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις ε, στον Ακόρνο Καραμπάχα. Η κλιμάκωση, η πρόσφατη κλιμάκωση επηρεάζει όχι μόνο τις δύο χώρες αλλά και όλη την περιοχή. Ελπίζω ότι η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και θα επιλέξουν μια ειρηνική επίλυση των, ε, της σύγκρουσης. Η σύγκρουση αυτή δεν μπορεί να επιληθεί εάν δεν υπάρχει ε, οικοδόμηση εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές και κοινοβουλευτική συνέλευση, η ισότιμη κοινοβουλευτική συνέλευση Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης ε, και των χωρών αυτών επιτρέπει να υπάρχει μια επαφή, να διατηρείται αυτή η επαφή ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν. Και ελπίζω όμως ότι δεν θα είναι αυτή η μόνη βοήθεια για την επίλυση της, του προβλήματος στην Αγκόρνο Καραμπάχ. υποστηρίζω μια πιο ε, έντονη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες ε, επίλυσης του προβλήματος. Ε, θα, προφανώς θα πρέπει να παραβιαστούν και οι αρχές της αυτοδιάθεσης των λαών και της διασφάλισης της εθνικής επικράτειας. Ελπίζω ότι οι αρχές αυτές, ο σεβασμός των αρχών αυτών Ε, θα βοηθήσουν ε, τις δύο αυτές χώρες να προχωρήσουν ε, στην ανάληψη των απαραίτητων βημάτων που θα είναι προς όφελος όχι μονάχα των, λαών αυτών αλλά και όλης της περιοχής. Συνάδελφος, ο πρόεδρος, συγγνώμη. Θα ήθελα να περιορίσουν οι συνάδελφοι που ζήτησαν τον λόγο τις παρεμβάσεις στα τρία λεπτά. Τον λόγο τον έχει ο αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα πολωνικά. Ένας ε, ομιλητής στο τέλος της ε, Παρέμβασή του είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός από τα τεθωρακισμένα, εκτός από τους ελεύθερους σκοπευτές κτλ. θα πρέπει να επιτρέψουμε την επαφή ανάμεσα στους πολίτες, ανάμεσα στη κοινωνία αν θέλετε, του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Αυτή είναι μια πτυχή την οποία δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε. Επίσης ε, θα ήθελα να κάνω ένα, μια ερώτηση για το κατά πόσον υπάρχει μια πολιτική συζήτηση και στις δύο χώρες για, την, για θέματα εμπιστοσύνης, αν θέλετε, αμοιβαίας εμπιστοσύνης. ασχολούνται, τους απασχολεί μάλλον το θέμα της έλλειψης επαφής ε, της δύο αυτές χώρες. Η κυρία Νικολάη, άλλη αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω ρουμανικά, γιατί είναι ευαίσθητο το θέμα, βλέπω πολύ κοινό και θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένη και πιο σαφής. Νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να χαιρετήσουμε αυτή την προσέγγιση που ήταν ε, πραγματικά αντικειμενική της ε, πραγματογνωμοσύνης αυτής, αυτής της διαδικασίας από πλευράς εμπειρογνωμόνων και πολιτικών που δέχονται τη μία ή την άλλη πτυχή του θέματος. Θα πρέπει να εξεύρουμε και απάντηση στο ερώτημα του Λένιν. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, τι πρέπει να γίνει. Στη συνέχεια, μετά το Λένιν, είχαμε το Στάλιν, ο οποίος ανέτρεψε και την τάξη πραγμάτων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την απτή πραγματικότητα δεν θα πρέπει να ξαναζήσει το παρελθόν του αυτός ο λαός. Θα πρέπει να εξεύρουμε μία λύση. Εάν θέλουμε να εξεύρουμε μία λύση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πόσο μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για χώρες οι οποίες βεβαίως δεν είναι γείτονες χώρες, αλλά μας ενδιαφέρει η κατάσταση του Καυκάσου, όπως μας ενδιαφέρει και η Γεωργία και ας μην είναι γειτονική χώρα. Εάν θέλουμε να εξεύρουμε μία ε, λύση, θεωρώ ότι θα πρέπει να εξευρεθεί μία λύση μέσα στα πλαίσια της ομάδας του Μίνσκ. Αν και ποτέ δεν έχει συνέλθει ομάδα στο Μίνσκ, διότι είναι μία δυσπρόσιτη περιοχή για ευνόητους λόγους. Ξέχουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, μεγάλα προβλήματα ορατότητας για την διεθνή κοινότητα η οποία δεν μπορεί να δράσει άμεσα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η κατάσταση ασφάλειας στο Νότιο κάφκας όπως μας ενδιαφέρει και στην Κεντρική Ασία. Έχουμε να κάνουμε με δύο παίκτες και την συμμετοχή της Ρωσίας και του Ιράν. Οι χώρες αυτές βρίσκονται πολύ κοντά, δίπλα στην Αρμενία. Υπάρχει βεβαίως και ο ιδιαίτερα ε, επίμαχος λόγος του Ιράν και του Ισραήλ. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε έναν παρεμπίπτοντα πόλεμο, έναν τυχαίο πόλεμο, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποσοβηθεί το Κοινοβούλιο έλαβε θέση με το ψήφισμα του 2010. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δείξει ενδιαφέρον σε αυτή την έφλεκτη ζώνη, θα πρέπει να ενδιαφερθεί για τα σύνορα αυτών των χωρών, γιατί ο Κάυκασος έδωσε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει θέση ως προς θέματα ε, παροχής ενεργειακών πηγών. Θα πρέπει να έχουμε μία ενεργό θέση, όπως κάναμε και στα Βαλκάνια. Δηλαδή ένα σύμφωνο σταθερότητας για τον Κάφκασο που να περιλαμβάνει και τη Γεωργία και το Αζερβαϊτζάν. Βεβαίως, οι αρχές της Μαδρίτης είναι ύψης της σημασίας. Θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή τη συζήτηση, την οποία θεωρώ ενδιαφέρουσα και άκρος αμερόληπτη. Euh, ευχαριστώ, κύριος Παλαισκής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτές τις τόσο συνεκτικές παρουσιάσεις. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις, κάποιες, κάποιοι πολιτικοί ηγέτες στον Πακού ή στο Ερεβάν. Ε, δεν φαντάζομαι ότι θα αλλάξει το καθεστώς στον Πακού, αλλά τέλος πάντων κάποιοι ηγέτες ή κάποια κόμματα τα οποία θα είναι διατεθειμένα να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Υπάρχουν τέτοια άτομα. Και δεύτερη ερώτηση. Αναφέρατε την Ρωσία, την Τουρκία, τις περιφερειακές δυνάμεις δηλαδή. Τι γίνεται όμως με τις παγκόσμιες δυνάμεις, με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Κίνα. Πώς προσεγγίζουν ε, την σύγκρουση αυτή, οι δύο αυτές δυνάμεις, συμπίπτει η προσέγγιση τους ε, και με, την, με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διαφορές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταρόντου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία ερώτηση στον κύριο, προς τον κύριο Λεφόρο, στον ε, ειδικό απεσταλμένο. Είχα κάποιες προφορίες πρόσφατα που λέει ότι παρά τις, ε, τα όσα γίνονται στον Κόρνο Καραμπάκα, κάποιες χώρες, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Γερμανία κτλ. πουλάνε ε, στρατιωτικό πολεμικό υλικό στο Αζερβαϊτζάν, κυρίως. Εσείς, ε, σαν ειδικό αποσταλμένος, ποια γνωμία έχετε. Αυτό δεν είναι μια παρέμβαση στον κώδικα συμπεριφοράς ε, που έχουν ε, υιοθετήσει τα κράτη-μέλη όσον αφορά την πώληση όπλων. Και εμείς σαν Επιτροπή του Κοινοβουλίου μήπως θα πρέπει να απευθυνθούμε στον ΟΑΣΕ και να του ζητήσουμε να μεταφέρει την, ε, την έδρα του από το Μίνσκ ε, λόγω των προβλημάτων ε, που υπάρχουν για την σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριο Στάνοκ, πολλά έχουν λεχθεί, καταρχάς σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κάμπερνακ. Πριν από πέντε χρόνια στην έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική γυτνίασης. Ε, είχα πει ότι ήλπιζα ότι τα πράγματα θα είχαν ε, εξελιχθεί. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, ακόμα βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Υπάρχει κλιμάκωση των, των εξελίξεων. Είχαμε τον, θάνατο 10 στρατιωτών. πολλά λέγονται ε, για, την, ε, για τα προβλήματα δημοκρατίας σε κάποιες, στην, ε, στην, στην, στο Αζερβαϊτζάν και τα λοιπά και τα κυβερνητικά προβλήματα, όμως δεν, δεν ξέρω τι θα γίνει με, το, με τις εξελίξεις όσον αφορά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. τι μπορεί να κάνει η, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εάν γίνει κάτι, μπορεί και οι Αρμένοι και οι Ρώσοι να καταλάβουν ε, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάποιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δηληστήρια στην ε, Κασπία. Και αυτό θα ανέβαζε απότομα τις τιμές του πετρελαίου. Επίσης ε, μπορεί να υπάρξουν ε, απώλειες ζωή, ε, ζωής, θα υπάρχουν πρόσφυγες που θα έρθουν σε εμά και σε χώρες όπως η, Γαλλία παραδείγματος χάρη, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί αρμενικής καταγωγής Γάλλοι. Λοιπόν, άρα πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευθεί αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή και όντως υπάρχει κίνδυνος, διότι υπάρχει και αυτή ε, η ανίερη συμμαχία ανάμεσα στην Ρωσία, στην ε, Αρμενία και στο Ιράν για εναντίον της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν που φαίνεται να μπορεί να ε, επεκταθεί και στη Γεωργία αλλά μπορεί να μπουν και άλλοι παίκτες αν θέλετε και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια σύγκρουση. Μπορεί να είναι μια σύντομη σύγκρουση όπως αυτή ανάμεσα στην Ρωσία και στην Γεωργία ή να εξελιχθεί σε κάτι ευρύτερο. Ε, και θυμόσαστε τι είχε γίνει πριν από τρία χρόνια, τρία-τέσσερα χρόνια ανάμεσα στη Ρωσία και στην Γεωργία. Ε, είδατε πώς ε, αντιμετωπίστηκε. Τότε ε, το, το, το μυαλό μας το είχαμε στις Ολυμπιακούς Αγώνες και προφανώς δεν ασχολούμεθα με τον Κάφκασο και ξαφνικά ξέσπασε ένα πόλεμος πόλεμος εκεί, ευτυχώς που ήταν περιορισμένος. Αλλά ελπίζω ότι, ε, ε, φοβάμαι μάλλον, ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο τώρα θα είναι πολύ πιο διευρυμένο το θέμα. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που πήραν το λόγο, αλλά και τους προσκεκλημένους. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ αμερόληπτη παρουσίαση. Στο πλαίσιο αυτής της σύγκρουσης, νομίζω ότι την ίδια στάση θα έπρεπε και εμείς να έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια στάση ουδετερότητας και αμεροληψίας ώστε να εξευρεθεί μια, λέξη, μια λύση συγγνώμη, στο πλαίσιο ε, της ε, ομάδας Μίνσκ ε, εποφελεί και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να έχουμε μια τάση να παίρνουμε το μέρος του ενός ή του άλλου, αλλά νομίζω ότι όταν δεν μας αφορά κάτι απολύτως άμεσα, δεν υπάρχει λόγος να παίρνει κανείς το μέρος του ενός ή του άλλου Αντιθέτως πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε μία λύση προς όφελος των πληθυσμών, γιατί και οι δύο πληθυσμοί ε, έχουν πληγεί, υπάρχουν εκτοπιστέντες ε, και στις δύο πλευρές και στις δύο πλευρές υπάρχουν πρόσφυγες όταν κάποιος είναι πρόσφυγας από την περιοχή αυτή ε, βρίσκεται σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε φυσιολογική, τουλάχιστον ε, όχι βάσει ευρωπαϊκών, ε, βάσει προδιαγραφών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει η κατάσταση δεν είναι απλή. Και πρέπει να πούμε στις κυβερνήσεις μας ότι πρέπει βέβαια να πάρουν τις αποστάσεις τους σε σχέση με οποιοδήποτε πρόγραμμα ε, βίας, γιατί ποιος θα ε, υποφεληθεί από όλα αυτά, ο μεγάλος γείτονας του Βορρά, η Ρωσία, ο οποίος μάλιστα θα παρουσιαστεί και όσο μεγάλος συνενευτής της ε, ε, όλης διαδικασίας, λέγοντας ότι ορίστε, ε, έκανα τις δύο χώρες ε, να συμφωνήσουν, αποκαθιστώντας τη ζώνη επιρροής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα επιθυμούσαν και οι δύο πλευρές, που θέλουν από μόνες τους να βρουν μια ειρηνική λύση. Βέβαια, η αναζήτηση αυτής της λύσης είναι δύσκολη. θα διευκολυνθεί από πλευράς Αζερβαϊτζάν αν όλος αυτός ο πλούτος που έχει το Αζερβαϊτζάν χρησιμοποιεί το για να ε, δημιουργηθεί μια πραγματικά ανοιχτή και διαφανής δημοκρατία τόσο πολύ ε, θελκτική που ο πληθυσμός του Ναγκόρνο Καραμπάχ θα έλεγε «Μα τι καταπληκτική χώρα, ε, πλούσια, ε, ευημερούσα χώρα με τόσο καλές κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης». Εκεί θα θέλαμε να ανήκουμε όμως, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Και πολύ δρόμο έχουμε ακόμη μπροστά μπροστά μέχρι να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τι μας μένει λοιπόν σε μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε. Μπορούμε, νομίζω, να προβλέψουμε τη δυνατότητα επιστροφή των προσφύγων και από τις δύο πλευρές. Αυτός είναι, είναι μια κατεύθυνση προς την ειρηνευτική διαδικασία είναι νομίζω από τα βασικά ζητήματα που μπορούμε να κάνουμε. Κυρία Κοπά. Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες για όλα τα ενδιαφέροντα σχόλια. Δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, η εντύπωση που έχουμε είναι ότι και τα δύο μέρη ε, είναι, φαίνεται ότι είναι ε, ικανοποιημένα με το status quo, διότι οι Αρμένοι δεν θέλουν να, να δώσουν ε, εδάφη τα οποία είχαν πάρει με τον προηγούμενο πόλεμο και οι Αζέρι θέλουν να να κάνουν κάτι μέχρι ότου αλλάξει η κατάσταση και είναι προς όφελός τους. Και η ερώτηση που κάνω είναι ποιο είναι ε, ποιο είναι το όπλο αν θέλετε, ποιος είναι, τι μπορούμε να ασκήσουμε σαν πίεση σε αυτές τις δύο χώρες. Τώρα, προς τον κύριο Λεφόρ μια ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με τη δήλωση του κύριου Έμπερχαρτ που λέει ότι είμαστε κοντά σε έναν ε, διευρυμένο πόλεμο. Αυτό το πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέγγελ. Όλοι μπαίνουν στον πειρασμό να πούνε κάτι παραπάνω ε, από τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας στην Επιτροπή για αυτό το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεκίνησε από τον ψυχρό πόλεμο, από την περίοδο του ψυχρού πολέμου και θα πρέπει να συνεισφέρουμε στην ανέβρεση μιας ε, λύσης ε, τώρα. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα βέβαια. Πολλές φορές προσπαθούμε να ισορροπήσουμε την κατάσταση χωρίς να υπάρχει ζυγαριά. Διότι εδώ έχουμε μια χώρα της οποίας το 60% σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δώσανε ε, έχει καταληφθεί και έχουμε ένα άλλο κράτος το οποίο έχει καταλάβει επικράτη άλλης χώρας και ε, εποφελείται κιόλας και από κάποια πλεονεκτήματα τα οποία εμείς σαν διεθνή κοινότητα δεν θα έπρεπε να επιτρέπουμε. Λοιπόν, εμείς πρέπει να επιβάλλουμε τον σεβασμό του Διεθνού δικαίου. Ένα πράγμα. Αυτό. Δεύτερον, είναι επικοδομητικό και θετικό το ότι προσπαθούμε να ε, απλώσουμε το χέρι και στις δύο χώρες σαν εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω αυτό να επιβάλλουμε την ανάγκη για αυτές οι δύο χώρες να βρουν μια συμβιβαστική λύση και να βρουν να βρούνε μια λύση γενικότερα που να είναι προς όφελος των πολιτών των δύο χωρών. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Και θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλα τα εργαλεία όπως παραδείγματο χάρη επαφές ε, μεταξύ των, ε, της κοινωνίας, ε, μεταξύ των πολιτών, διαρθρωμένες επαφές έτσι ώστε ο κόσμος να έρθει, κοντήτε, να έρθει πιο κοντά. Όμως αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει και δεν θα πρέπει να στέλνει δηλαδή ένα, το λάθος μήνυμα στην Αρμενία ότι δεχόμαστε το status quo, όπου τώρα με τη βοήθεια των Ρώσων και των ρωσικών όπλων η Αρμενία προσπαθεί να νομοποιήσει μία κατάληψη. Αυτό δεν είναι σωστό και θα πρέπει να το ξέρουν οι Αρμένοι. Merci, Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Uh, while following the talks Παρακολουθώ τη συζήτηση για τον Αγκόρνο Καραμπάχ εδώ και πολλά χρόνια και πραγματικά δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος ε, με την ε, εξέλιξη της κατάστασης αλλά και με την αξιολόγησή της ε, Τι χρειαζόμαστε καταρχάς. Νομίζω ότι πρέπει να καθαρίσουμε, να είναι ξεκάθαρο και το μυαλό μας αλλά και το λεξιλόγιό μας ε, όταν ε, ε, μιλάμε για αυτό το θέμα. Ας βρούμε τέλος πάντων έναν τρόπο να μιλήσουμε καθαρά. το line of contact ας πούμε. Υπάρχουν ε, ειρηνευτικές ε, ε, διαδικασίες που να έχουν ξεκινήσει. Αν όχι δεν είναι line of contact αλλά είναι line of shooting. Δεν είναι δηλαδή γραμμή επαφής, είναι γραμμή πυροβολισμών. Και τι γίνεται δηλαδή... Ε, για ποιο λόγο εξακολουθούν να υπάρχουν όλες αυτές ε, ε, οι χαμένες ζωές και τι κάνει γι' αυτό η ομάδα του Μίνσκ. πόσο καιρό θα συνεχίσει αυτό, γιατί και ο κύριος Έμπερχαρτ το είπε καθαρά, η... λέμε ότι η Ρωσία φταίει για αυτήν τη στρατιωτική βία. Και όταν φτάνουμε στη Ρωσία, ε, τότε αρχίζουμε να μιλάμε πραγματικά. Γιατί ε, η Ρωσία θα το ήθελε αυτό, γιατί πραγματικά θα ήταν μια ευκαιρία για τη Ρωσία να παρέμβει όπως έγινε και στη Γεωργία και ε, θα ήταν ένας τρόπος να ελέγξει και το Αζερβαϊτζάν, γιατί την Αρμενία την ελέγχει ήδη. Οπότε η Ρωσία παρουσιάζεται σαν ειρηνευτής σε αυτή την περίπτωση. Α συγκρίνουμε και του προπολογισμού του στρατιωτικού, ε, ε, συγκρίνουμε τη Αρμενία με το Αζερβαϊτζάν, α συγκρίνουμε το Αζερβαϊτζάν με τη Ρωσία καλύτερα και τότε θα δούμε την ευρύτερη ε, εικόνα. Η Αρμενία λέει ότι δεν θέλει καμία παραχώρηση. Αν δεν υπάρξουν όμως παραχωρήσεις, ε, θα υπάρξει τελικά πόλεμος. Επίσης μιλάμε για συγκρούσεις μεταξύ και των δύο πλευρών. Σε ποια πλευρά όμως είναι η Ρωσία, τι εννοείται μεταξύ δύο πλευρών. Γιατί είναι ένα προτεκτοράτο της Ρωσίας η Αρμενία. Άρα γιατί μιλάμε μόνο για δύο πλευρές. Επίσης λέμε για ένα, μιλάμε για ε, διαφιλονικούμενο, ε, για μια διαφιλονικούμενη περιοχή. Ε, όχι, είναι κατεχόμενη περιοχή, δεν είναι απλώς ε, διαφιλονικούμενη. Εφόσον υπάρχει ψήφισμα απόσυρσης από τα κατεχόμενα γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ε, είναι κατεχόμενη αυτή η περιοχή. Να μιλάμε λοιπόν καθαρά. Περί αυτού πρόκειται. Να μην ε, μπερδευόμαστε μεταξύ μας. Έτσι που μπερδευόμαστε δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τίποτα, ούτε να λύσουμε την ε, σύγκρουση, να επιλύσουμε τη σύγκρουση. Παρακαλώ, αν είναι, να αρκείστε στα τρία λεπτά, αλλιώς δεν θα πρόκειται να γίνει συζήτηση. Ο κύριο Κυρίλοφ, θα ήθελα να επικεντρωθώ στα εξής. Σύντομα. Νομίζω ότι και κάποιοι από του προσκεκλημένου μα το είπαν ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο προς την ειρηνευτική ε, κατεύθυνση, ναι, απολύτως, αλλά αυτό σημαίνει αναθεώρηση και της στρατηγικής και με αυτό συμφωνώ. Ένα ακόμη ερώτημα που ετέθη είναι οι δύο πλευρές ε, της σύγκρουσης θέλουν μια πιο ενεργό συμμετοχή. Εγώ έχω την εντύπωση ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυριαρχεί αυτή η εντύπωση ότι θα έπρεπε να εμπλακούμε. Για ποιο λόγο? Εμείς δεν είχαμε εμπλακεί ιδιαίτερα ε, στην κρίση με τη Γεωργία, όμως έπρεπε να αντιδράσουμε και ε, μάλιστα με ε, μεγάλο τίμημα, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις εμπλεκόμενες χώρες. Αν ρωτήσουμε αυτές τις δύο χώρες, και αυτό είναι το ερώτημα που θα ήθελα να ε, θέσω προς τον κύριο Λεφόρ, θα αντιδράσουν θετικά στην πιο ενεργό ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη σας και οι δύο χώρες ε, συμφωνούν με αυτήν την, ε, κατά τη γνώμη μου, πολύ κανονική κατάσταση βάσει της οποίας εμείς θα έπρεπε να έχουμε ανεφόρον πρόσβαση πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε αυτό το πράγμα αν θέλουμε μια ειρηνική επίλυση σύντομα ποιος θα είναι ο ρόλος μας ε, σε αυτή τη διαδικασία την ειρηνευτική. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει η Αρμενία, εντάξει εμείς να αποσυρθούμε αλλά έχουμε εγγυήσει ασφάλειας, μήπως θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα με τις χώρες αυτές ανοιχτά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα ζητήματα από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Ο κύριος Κοβάτσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ καθόλου τη διάρκεια της συζήτησης, αλλά δυστυχώς ε, είχα ε, μία άλλη υποχρέωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί το Ναμπόρνο Καραμπάχ δεν είναι μόνο ένα, μια παγωμένη σύγκρουση, αλλά ε, ε εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ε, θανατηφόρα περιστατικά ε, στην ε, γραμμή επαφής και αυτό είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γνωρίζουμε προς ποιας πλευράς το όφελος είναι αυτή η κλιμάκωση της σύγκρουσης, είναι πιο επωφελής για την Αρμενία, το να μην βρεθεί μια λύση ε, σωστή ή είναι προς όφελος του Αζερβαϊτζάν. Νομίζω ότι πρέπει να διερευνήσουμε, να παρατηρήσουμε ποιος, ποια από τις δύο πλευρές έχει περισσότερο συμφέρον να εξευρεθεί μια λύση αμέσως, τέλος πάντων βραχυπρόθεσμα, ε, και ποιος έχει συμφέρον ε, να διατηρηθεί το status quo και να μην σκεφτόμαστε μόνο την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, αλλά και τις γύρω χώρες, τις γειτονικές χώρες. Και τότε βέβαια θα έχουμε μια πολύ σαφέστερη εικόνα για το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν θα έπρεπε να ακολουθήσουν ε, τις ε, συστάσεις του Κοινοβουλίου ε, για την ε, απομάκρυνση των ελεύθερων σκοπευτών. Δεν ξέρω γιατί δεν συμβαίνει αυτό και για ποιο λόγο. Ναι, ναι, λένε και οι δύο πλευρές, ε, τουλάχιστον στα λόγια και λένε ότι επί τη αρχής δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά τελικά στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ομάδα Μίνσκ και όλοι τέλο πάντων οι διεθνεί εμπλεκόμενοι πρέπει να αναλάβουν δράση. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αν όντως κάποιοι στρατιώτες ε, δημιουργήσουν τελικά μία κλιμάκωση της ε, σύγκρουσης ε, και τελικά αυτή η λανθάνουσα τέλος πάντων σύγκρουση τελικά εξελιχθεί σε πόλεμο κανονικά δημοκρατικές χώρες ε, δεν αρχίζουν πόλεμο μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εμείς ε, να επενδύσουμε στη δημοκρατία, στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις δύο χώρες ε, σε μια καλή κοινοβουλευτική δημοκρατία, να συζητήσουμε και με τα δύο κοινοβούλια, να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας, επαφές μας με την κοινωνία των πολιτών και στις δύο πλευρές, γιατί η πρόληψη του πολέμου και της ασφάλειας στην περιοχή έχει άμεση σχέση με το επίπεδο της δημοκρατίας ε, και έχει και επίδραση και στις υπόλοιπες ε, ε, χώρες της περιοχής, συγκεκριμένα κυρίως στην Αρμενία και τον Αζερβαϊτζάν. Και το Αζερβαϊτζάν. Η πρόληψη των συγκρούσεων για μένα έχει άμεση σχέση με το επίπεδο της δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, στις δύο χώρες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Επίσης, τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πάρα πολύ ανησυχώ και είμαι και πάρα πολύ απογοητευμένη. Εγώ είμαι ε, Σουηδή Ευρωβουλευτή, αλλά ξέρετε ότι είμαι και πρόσφυγας ε, από ε, την Βοσνία. Για μένα είναι déjà vu όλο αυτό που συμβαίνει. Νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Ε, και μιλάω για τη Ρεπούμπλικα Σύρψκα από την οποία προέρχομαι εγώ. Όταν υπάρχουν κατεχόμενα, η κόσμος φεύγει, τότε ε, ε, σιγά σιγά μειώνεται ο αριθμός των ατόμων, ε, ε, τελικά τα πράγματα βέβαια διορθώνονται. τώρα έχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση η περιοχή από την οποία έρχομαι εγώ. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνει ο κόσμος στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Υπάρχει όμως και το θέμα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και του πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Εμείς λέμε ότι είναι μια σύγκρουση μεταξύ δύο χωρών, όμως είναι μια κατοχή, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πάμε πίσω στο ε, πώς ξεκίνησαν όλα. Ζητάμε από τους δύο να κάνουν μια ε, προσπάθεια όμως ποτέ δεν είδαμε τελικά ποιο είχε δίκιο και ποιο είχε άδικο και ως πολιτικοί πρέπει να έχουμε το στένος να πούμε ότι κάτι είναι λάθος, πρέπει να έχουμε το στένος να πούμε ότι πρόκειται για μια κατοχή. Εγώ συμφωνώ να επιστρέψουν οι πρόσφυγες, συμφωνώ με την αυτοδιάθεση, όμως πρώτα πρέπει να σταματήσει η κατοχή και τότε να γυρίσουν οι πρόσφυγες. Τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια επίλυση. Μετά από όλα αυτά, κάποιος είπε προηγουμένως από το πάνελ, ε, μίλησε για το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ειρήνης της Στοκχόλμης και λέει ότι, λέει ότι πώς ε, ποια είναι οι στρατιωτικές δαπάνες για το στρατιωτικό εξοπλισμό του Αζερμπαϊτζάν. Εγώ είμαι Σουηδέζα, διαβάζω τα ίδια πράγματα. Ε, αν πάτε στην, στο site τους θα δείτε ότι αν δεν υπάρχουν τα σωστά νούμερα για την ε, ε, Ρουμανία, για παράδειγμα, είναι γιατί δεν δίνονται τα σωστά στοιχεία ε, στην δημοσιότητα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε. Εγώ είμαι υπέρ της κοινωνίας των πολιτών και την συνεργασία ε, με την κοινωνία των πολιτών, αλλά τι κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνουμε τα μάτια μας, έχουμε στρατιωτική παρέλαση στον Αγκόρνο Καραμπάχα, ε, έδειξαν, έκαναν επίδειξη των όπλων που έχουν και αυτό είναι μια, ένα σαφές μήνυμα και προς το Αζερβαϊτζάν και προς εμάς. Κύριε Λεφόρ, αντέδρασε κανείς σε αυτό, Είπε κανείς στην Αρμενία ότι δεν πρόκειται να υπάρξει περισσότερη ειρήνη ε, με τέτοια πράγματα. Εγώ θα ρωτήσω και την ε, κυρία Άστον απευθείας για το θέμα αυτό. Βλέπω ότι η συζήτηση είναι ιδιαίτερα ζωηρή. Νομίζω ότι εκφράστηκαν όλοι. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη θα ήθελα οι τρεις εμπειρογνώμονες και ο κύριος Λεφόρ να συνοψίσουν. Έχετε πέντε λεπτά ο καθένας. Θα απαντήσετε ως προς το σκέλος ή τα σκέλη που σας ενδιαφέρουν και θα ε, συνοψίσει και ο κύριος Λεφόρ. Η κυρία Τζέρμαν. Ευχαριστώ. Έγινε λόγος για, τους, για εξωτερικούς παράγοντες και φορείς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επιληθεί αυτή η εμπόλεμη κατάσταση χωρίς να λάβουμε υπόψη τον ρόλο των φορέων εκτός από την Αρμενία και την, το Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή να δούμε το Ιράν, την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία για να προωθηθεί η σταθερότητα ή αστάθεια, δεν ξέρω. Ε, δεν μπορεί να επιληθεί αυτή η διαφορά χωρίς να συμμετέχουν όλοι. Ε, έγινε λόγος για ένα σύμφωνο σταθερότητας και καταβλήθησαν πολλές προσπάθειες για να συσταθεί ένα σύμφωνο σταθερότητας. Πρόσφατα είχαμε την ε, πρόταση της ε, Ρουσίας ε, το 2008 την πλατφόρμα ανάπτυξης και σταθερότητας του Καυκάσου, αλλά απέτυχαν όλες αυτές οι πλατφόρμες διότι απέκλεισαν συγκεκριμένες φο... συγκεκριμένους φορείς η Τουρκία απέκλεισε το Ιράν, για παράδειγμα. Και αν θέλουμε ένα τέτοιο σύμφωνο σταθερότητας, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όλους τους παράγοντες και φορείς που έχουν κάποιο ρόλο να διαδραματίσουν στον Κάφκασο. Ως προς τη σύνθεση της ομάδας Μίνσκ, η ομάδα Μίνσκ αντιμετωπίζει προβλήματα και οι συμπροεδρίες έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Αλλά θα πρέπει να φτάσουμε στην επίλυση του, της διαφοράς γενικότερα και όχι να μιλάμε για νέα σύνθεση της ομάδας του Μίνσκ. Κάποιος αναφέρθηκε στο status quo έγινε μια δημοσκόπηση το 10 νομίζω στην Αρμενία. Πάνω από το 40% του πληθυσμού της ε, Αρμενίας που είναι 3 εκατομμύρια θα έφευγαν από τη χώρα αν μπορούσαν διότι οι οικονομικές προπτικές δεν είναι καλές. Η οικονομία πλήττεται από οικονομική κρίση και γι' αυτό ίσως το status quo κάτι υπηρετεί. Πλήττονται οι πληθυσμοί από αυτό, μην το ξεχνάμε. Οι άλλοι εμπειρογνώμονες θα μιλήσουν περισσότερο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά νομίζω ότι ε, θα ήταν σκόπιμο ε, να δώσω τα δύο μου λεπτά στους άλλους ομιλητές, γιατί νομίζω θα έχουν να πούν περισσότερα για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι, και ρωτήσατε αν οι κοινωνίες σε αυτές τις δύο χώρες είναι όριμες για την αλλαγή και αν μπορούν να επηρεάσουν. Στο τέλος τη δεκαετίας του 90, η ελίτ και από τις δύο χώρες λέγαμε ότι ήταν έτοιμες για συμβιβασμό. Οι κοινωνίες δεν ήτανε. Τα τελευταία 10 και 15 χρόνια όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μετακίνηση στην πολιτική, στις πολιτικές ελίτ της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν. Γίνανε γεράκια και ε, είναι πιο φανατικοί αν θέλετε και βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις και των δύο χωρών κάνουν ό,τι πρέπει για να μην είναι οι κοινωνίες ε, έτοιμες να δεχτούν συμβιβασμό. Ακού, ακούστηκε και μία ερώτηση για τη θέση των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατάνε χαμηλό προφίλ και κάπως και σχετικά ισορροπημένη θέση τους για δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ότι υπάρχει ένα ισχυρό αρμενικό λόμπι στις πολιτείες και επηρεάζει το Κογκρέσο και το Κογκρέσο επιβάλλει περιορισμούς στην πώληση όπλων στο Αζερβαϊτζάν. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Αζερβαϊτζάν παίζει και ένα σημαντικό ρόλο στον ε, τομέα της ενέργειας στην γεωπολιτική της ενέργειας. Και κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι το Ιράν, το Αζερβαϊτζάν είναι ένας ισχυρός παράγοντας στην περιοχή. Τώρα για την Κίνα, το, ενδιαφέρον της Κίνας είναι περιορισμένο επί του παρόντος και η Κίνα δεν έχει εμπλακεί ενεργά. Ενδεχόμενα σε 5, 10, 15 χρόνια είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν τα πράγματα όταν οι κινέζικες εταιρείε ε, θα κατασκευάσουν τον ε, αγωγό που θα περνάει από, την, τον Κάφκασο. Όχι όμως τον αγωγό της, ε, του Καυκάσου όπως τον θέλουμε εμείς που θα πηγαίνει προς την Δύση, αλλά θα, τον αγωγό που θα περνάει από τον Κάφκασο και θα πηγαίνει και θα στέλνει το πετρέλαιο του Αζερβαϊτζάν ανατολικά, στην Κίνα. Τώρα, για να διευκρινίσω τη θέση μου για το, ενδεχό, για το πώς βλέπω να εξελίσσεται και ή αν θα υπάρξει σύγκρουση, να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για το Αζερβαϊτζάν να ξεκινήσει ένα πλήρη πόλεμο. Αλλά ο η απειλή ενός τέτοιου πολέμου αυξάνεται και όντως σε τρία με πέντε χρόνια φοβάμαι, φοβάμαι ότι ενδεχόμενα θα συμβεί. Τελευταίο ερώτημα για αυτή την αναλογία των στρατιωτικών δαπανών, ε, το ποσοστό στρατιωτικών δαπανών στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν. Στην παρουσίαση μου είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε τις στρατιωτικές δαπάνες γιατί οι προϋπολογισμοί είναι, ε, ε, εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, σε πάρα πολλά κονδύλια του, κρατικού προπολογισμού υπάρχουν στρατηγικές δαπάνες, έχουν ενσωματωθεί στρατηγικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι το Αζερβαϊτζάν... Μάλλον μπορούμε να πούμε ότι το Αζερβαϊτζάν έχει χρήματα και μπορεί να δαπανίσει ε, πολλά για τις στρατιωτικές δαπάνες, για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Ενώ η Αρμενία λόγω της οικονομικής κατάστασης δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πρόεδρε, υπήρξε μια ερώτηση για το κατά πόσον υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες που είναι πιο μετριοπαθείς από κάποιους άλλους. Από εκεί θα ξεκινήσω. Πριν από 1,5 χρόνο κάναμε μια έρευνα ε, σε 46 πολιτικά κόμματα στην Αρμενία και 23 στο Αζερβαϊτζάν. Του ζητήσαμε συγκεκριμένα να μας πούνε τις απόψεις τους για το πρόβλημα του Καραμπάχ. Η έρευνα αυτή δείχνει ότι και στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν υπάρχει μια γενικότερη συνένεση για το πώς βλέπουν να εξελίσσονται τα πράγματα και αυτό έπρεπε να το περιμένουμε. Διότι αν κάποιος ο πολιτικός ε, αποκλίνει από την πολύ από την γενική εθνική γραμμή, αυτό θα σημαίνει την πολιτική του αυτοκτονία. Όμως, από την άλλη πλευρά, αν δείτε τις απαντήσεις που έδωσαν πολλοί στις ερωτήσεις μας, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες αποχρώσεις. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να, χτίσουμε αυτές τις αποχρώσεις, για να ενθαρρύνουμε τις συζητήσεις, πιστεύω. Αυτή είναι μια συζήτηση που οι πολιτικοί των χωρών αυτών πρέπει να κάνουν μόνοι τους. Εμείς όμως μπορούμε να υποστηρίξουμε την διαδικασία αυτή. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τον απαραίτητο χώρο, το πλαίσιο που θα λάβουν χώρα αυτές οι συζητήσεις. Και χρήσιμα πράγματα θα βγουν από αυτή τη συζήτηση, διότι από τη μία πλευρά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα πιο σκληροπρινικοί από τις κυβερνήσεις, όμως υπάρχουν και κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις. Πιστεύω πρέπει να ακούγονται περισσότερο. Και επίσης υπάρχει αυτή η ερώτηση με την συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό των κοινωνιών. Ένα από τα πράγματα στα οποία μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δημιουργήσει ασφαλείς χώρους συζήτησης και στο εσωτερικό των χωρών αλλά και ανάμεσα στις χώρες και στις κοινότητες και πιστεύω ότι θα πρέπει να τα βάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και θα ήθελα να κάνω μια προειδοποίηση, αν θέλετε, όχι γιατί δεν το έχουν πει και στο παρελθόν. Για 15 χρόνια συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις και ξέρω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Όμως, ένα από τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν ήταν ότι υπήρχε ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα αυτά οποία γινόταν ε, στην κοινωνία από τη μια και στην ε, ειρηνευτική διαδικασία από την άλλη. Διότι η ειρηνευτική διαδικασία αυτή δεν ήταν ευαίσθητη, αν θέλετε, στα όσα γινόντουσαν γύρω της, ε, δεν ήταν ευαίσθητη στο περιβάλλον. Και από την εμπειρία του παρελθόντος νομίζω ότι έχουμε διδαχτεί. Και εδώ μπορούσε να ήταν χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε να κάνει πράγματα τα οποία να βοηθάνε την όλη διαδικασία και έχουμε μέσω πίεση, ε, πρόεδρε. Άκουσα ότι η διεθνή κοινότητα δεν έχει ε, όπλο πίεση. Και όμω έχουμε, διότι όλε αυτέ οι κοινωνίε βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν έναν χώρο που του καταλαβαίνουν, από τον οποίο μπορούν να αντλήσουν νέε ιδέε ε, και βλέπουν ότι αυτέ είναι κοινωνίε που θα θέλουν. Κοινωνίες με τις οποίες θα θέλουν να μοιάσουν και στις χώρες τους. δεν μας βλέπουν μόνο σαν χρήματα αν θέλετε, ε, μας βλέπουν και σαν πρότυπα. Και αυτό πρέπει να το ε, χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να υποφεληθούμε από αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Λαντσμπέργκερ ότι η ορολογία που χρησιμοποιεί κάποιος ίσως να μην είναι ε, ιδιαίτερα κομψή. Λέγεται διαδικασία Μίνσκα. Κανείς δεν συναντήθηκε στο Μίνσκ. Η Λευκορωσία δεν έχει να κάνει τίποτα με την ιστορία αυτή και η γραμμή επαφής. Δεν υπάρχει η επαφή, αλλά μιλάμε για επαφές ανάμεσα στους στρατιωτικούς. Δηλαδή υπάρχει μια κάποια ορολογία την οποία χρησιμοποιούμε ε, και την οποία σιγά σιγά ίσως θα πρέπει να τροποποιήσουμε όσο, το, όσο εξελίσσεται το πρόβλημα αυτό. Τώρα, πρέπει να κρατήσουμε σε, σε πρωταρχικό, σε, σε βασική θέση, σαν θέση προτεραιότητα στην επίλυση του, της διένεξης αυτής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πείσουμε τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών να αντιμετωπίσουν την σύγκρουση αυτή από μια διαφορετική σκοπιά από αυτή που την βλέπανε στο παρελθόν. Για τη Ρωσία τώρα κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με όσα ακούστηκαν εδώ για τον αμφιλεγόμενο ρόλο της Ρωσίας που είναι στρατιωτικός σύμμαχος ε, της μίας πλευράς ε, και ε, συμμετέχει με έναν άλλο τρόπο στην διαδικασία επίλυσης του, της σύγκρουσης. Όμως ο ρόλος της Ευρώπης και η θέση της Ευρώπης είναι να επιτρέψει στη Ρωσία να συμμετέχει στην διαδικασία και να είναι πιο επικοδομητική στην επίλυση του προβλήματος. Η ιδέα να έχουμε ένα μνημόνιο σταθερότητας του Καυκάσου ή μια συνθήκη σταθερότητας του Καυκάσου που το έχει συζητήσει και το κοινοβουλευτικό και ψήφισμα πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε και πρέπει να το προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Όχι γιατί πρόκειται να συμβεί άμεσα, αλλά γιατί πρέπει να συμβεί κάποια στιγμή πριν επιληθεί πλήρως το, το πρόβλημα αυτό, η σύγκρουση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω πολύ γρήγορα, ε, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ήταν κοινά σε όλε τι συζητήσει. Το ένα είναι αυτό που ανέφερε ο κύριο Στάνοκ, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα. Αυτό το σενάριο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε. Ε, και μπορεί να υλοποιηθεί, διότι αν τα πράγματα μείνουν ω έχει, αυτή είναι η φυσική εξέλιξη, όλη αυτή η απογοήτευση η οποία έχει συσσωρευτεί όλε αυτέ οι δύσκολε δυσκολίες, τα εσωτερικά προβλήματα της μιας της άλλης χώρας. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάνω στο τραπέζι και το οποίο δεν το βλέπουν ε, οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί ε, των, χωρών αυτών. Πραγματικά με εκπλήσει το γεγονός ε, το ότι οι πολιτικές ελίτ και των δύο χωρών ε, οδηγούνται από την εικόνα που είχαν για τον πόλεμο του 1994 με τα Καλάσνικοφ, με τα δεν ξέρω εγώ με τι όπλα. Ε, δεν λαμβάνουν υπόψη τους πλέον τις καταστροφικές συνέπειες των νέων όπλων που δεν αφήνουν κανένα καμία ζώνη ασφάλειας σε καμία χώρα. Και το πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο για τις δύο αυτές χώρες ε, ότι δεν θα, δεν θα υπάρχει ζώνη ασφάλειας, αλλά για όλο τον Κάφκασο. Τώρα, κάτι άλλο για το ρόλο της Ρωσίας. Είναι αλήθεια ότι η Ρωσία είναι και διαιτητής αλλά και, και παίκτη. Διότι ε, προσφέρει και πουλάει όπλα και στις δύο χώρες τα ίδια όπλα και στην Αρμενία και στο Αζερβα... Αζερβαϊτζάν. Και είναι μια δύναμη, αν θέλετε, που θέλει να ελέγχει την περιοχή σαν κληρονόμος της Σοβιετικής Ένωσης. Υπάρχουν οι προοπτικές του Σότσι βέβαια, υπάρχουν κάποια ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή και σε οικονομικό και σε γεωπολιτικό επίπεδο και τα συμφέροντα αυτά θα, διακυ... θα τεθούν σε κίνδυνο εάν υπάρχει μια, ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας στην περιοχή αυτή. Άρα το μήνυμα που πρέπει να σταλεί είναι ένα μήνυμα μετριοπάθειας. Τώρα, μπορούμε να διαρωτηθούμε εάν η Ρωσία έχει συμφέρον να διατηρηθεί αυτή η σύγκρουση χαμηλής όμως ε, ε, χαμηλής ε, έντασης. Δηλαδή όπως η Αρμενία να διατηρήσει έναν, μια απειλή πάνω στην, στο Αζερβαϊτζάν και να μπορεί με τον τρόπο αυτό η Ρωσία να ελέγχει όλο τον Κάφκασο και κυρίως την ε, Γεωργία. αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό της Ρωσίας του, της δεκαετίας του 90. δηλαδή να εξάγει μια ένταση σε κάποιο σημείο της περιοχής έτσι ώστε να μπορεί να επωφελείται ε, σε, σε ένα διεθνές επίπεδο. η Ρωσία προσπαθεί να προωθήσει τα συμφέροντά της από τη μια, αλλά θα πρέπει να προσπαθεί ταυτόχρονα να διατηρήσει κάποια σταθερότητα στην περιοχή. και ίσως ε, ε, και προς το συμφέρον της Ρωσίας είναι ε, να μην επιληθεί το πρόβλημα του Καραμπάκ, αλλά να φύγουμε και από το status quo. Τέλος πάντων, εμείς τώρα ποια είναι η θέση μας. Εμείς είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Αλλά δεν μπορούμε όμως να αντικαταστήσουμε εμείς την θέληση των, των δύο εμπλεκομένων. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε ενδεχόμενα, μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε την ειρήνη. Αυτή, αυτή μπορεί να την, να επιλέξουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι. Και συζήτηση, ερώτηση που έγινε προηγουμένως, να σας πω ότι δεν συζητάνε καθόλου για το θέμα αυτό, ούτε στην Αρμενία, ούτε στο Αζερβαϊτζάν. Όλοι ξέρουν τη διαδικασία της Μαδρίτης, αλλά την αγνοούν, δεν την συζητάει κανείς. Είναι θέμα ταμπού. Επομένως θα πρέπει για άλλη μια φορά να έχουμε κατά νου ποια είναι η προοπτική, μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη. υπάρχουν ε, σκαμπανεβάσματα, αν θέλετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Φυσικό είναι, θεωρώ. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα υπάρξει ειρήνη, όπως και στη Βόρεια Ιρλανδία, που θεωρούσαμε πριν από μερικά χρόνια ότι ήταν καταδικασμένη η κατάσταση. Θα υπάρξει όμως ειρήνη όταν οι δύο χώρες και οι δύο ηγεσίε συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτές τις δύο χώρε εάν δεν υπάρξει ένα συμβιβασμό δύσκολο και οδυνηρός. Ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει όμως. Και πρέπει αυτό να το προωθήσουμε εμεί αυτή την ευαισθητοποίηση των ηγετών των δύο χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή και για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες που προσήλθαν. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί Ελπίζω να μην, συμβεί, να μην έχουμε τίποτα πρόπτα το καλοκαίρι όπως συνέβη με τον Κάφκασο και παρά τη, τους κινδύνους που διατρέχουμε θα διακόψουμε για δύο λεπτά και θα ασχοληθούμε με τα ευρωπαϊκά συστήματα ραθιοπλογήσεις με δορυφόρο. S'il vous plaît, je demanderai personnes qui doivent quitter la salle. Παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν γιατί έχουμε ακόμη και άλλες εργασίες στην υποεπιτροπή μας. Merci. Et donc, le sujet... Ευχαριστώ πολύ. Σύστημα ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου, έγνος και γαλιλαίο. Γνωρίζετε ότι τα προγράμματα αυτά είναι πάρα πολύ δαπανηρά και ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τη χρηματοδότησή τους. Η Επιτροπή Ήτρε είναι ε, αρμόδια. Εμείς γνωμοδοτούμε απλώς. Ο κύριος Τέρο θα μας πει, θα μας κάνει τα σχόλιά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ θα μιλήσω φινλανδικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ε, εισηγητές και όλη την Επιτροπή για τα σχόλια. Ε, θα μπορούσα να υποστηρίξω τους περισσότερους. Μας ακούτε? Για ε, το σύστημα Galileo ε, έχουμε ε, βασικά προβλήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να έχουμε επεξηγήσεις ως προς την τροπολογία 17 δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να γίνει αυτή η μνήα. Θα ήθελα να μας εξηγήσει η κυρία Νικολάη τι σημαίνει, τι mutual ownership. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορεί να οριστεί εκ νέου αυτή η τροπολογία. Στο, στην τροπολογία ε, θα ήθελα κυρία Κόρμαϊ να καθίσει και να βάλει τα ακουστικά της. Την 25 γίνεται ένα σχόλιο σε σχέση με την κοινοποίηση στο Κοινοβούλιο εν χρόνο. Αυτό το εν χρόνο στην 25 δεν με πείθει. Στην τροπολογία 29 δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να γίνει μια νέα ε, διαμόρφωση και σύνταξη. Αυτό που προτείνεται να απαλληφθεί, μπορείτε να μας επεξηγήσετε γιατί πρέπει να απαλληφθεί. Ως προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν θα ήθελα να σχολιάσει τις 32 και 38, το τρίτο μέρος της 38. Να μας πει δηλαδή κατά πόσο αντικατοπτρίσουν την παρούσα κατάσταση μεταξύ Κομισιών και Συμβουλίου. Όπως σας είπα, οι τροπολογίες είναι πάρα πολύ καλές και από τότε που το συζητήσαμε πιστεύω ότι έχει επιτελεστεί η πρόοδος σε σχέση με την τελική εκδοχή της έκθεσης. Χρειαζόμαστε τροπολογίες συμβιβασμού και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πολύ καλή αυτή η νομοθέτηση. Ε, πολύ ευπρόσδεκτα όλα σας τα σχόλια. Θα δώσω το λόγο στους συντάκτες. κυρία Νικολάη. Κυρία Νικολάη. Έχετε κάτι να πείτε? Ε, μόνο μία επεξήγηση θα ήθελα να σας ε, δώσω. Η νομική κατάσταση, γιατί ποτέ δεν ετέθη το ζήτημα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό μιλάμε για το mutual ownership, τη δυνατότητα δηλαδή για όλους και τους πολίτες και τους στρατιωτικούς να μπορούν να τη χρησιμοποιούν. Εγώ είχα σκεφτεί ε, να κάνουμε τη συζήτηση και υπό αυτό το πρίσμα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, ε, συντάκτη της γνωμοδότησης. Νομίζω ότι θα προς τη σωστή κατεύθυνση ως προς την υποστήριξη της ε, χρήσης ε, του δορυφόρου και για πολιτικούς αλλά και για στρατιωτικούς σκοπούς. Προφανώς είναι προς όφελος των στρατιωτικών και πολιτικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση των συστημάτων αυτών ώστε να μπορεί να είναι στρατηγικός ανεξάρτητη. Όσον αφορά τώρα στις τροπολογίες, ε, δεν θα υπερασπιστώ τις δικές μου, αλλά έχω ένα ερώτημα. Υποστηρίζω όλες τις ε, τροπολογίες που έχουν να κάνουν ε, με, τους, ε, με το στρατιωτικό και πολιτικό δυναμικό ε, του συστήματος αυτού, αλλά όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως όχι μόνο σε αμυντικούς και στρατιωτικούς στόχους, αλλά και στις αποστολές το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας παραμένει εκρεμές. Οπότε καλύτερα να επικεντρωθούμε στις αποστολές και μιλάω για τις τροπολογίες 28 και 38 Θα ήθελα όμως να μου πείτε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα, κατά πόσο είναι φυκτό κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λίγο περισσότερες πληροφορίες πριν να τοποθετηθώ για τις τροπολογίες που μόλις ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόπα. Uh, Υπέβαλα 10 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής έτσι ώστε να δω ορισμένα θέματα ουσίας. Ιδιαίτερα στην αιτιολογική σκέψη σε σχέση με την φύση αυτού του εγγράφου για να υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν υπόψη περισσότερο αυτές οι συστάσεις από την Ήτρε. Δεν νομίζω ότι ήδη στο δεύτερο θέμα να μιλήσουμε για τη δετή φύση του Γαλιλαίου σε συνδυασμό το, του δικαιώματος των κρατών μελών το χρησιμοποιήσουν για λόγους άμυνας και ασφάλειας. Δεν θα πρέπει να γίνει δήλωση στην αρχή του κειμένου. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την σημασία του Γκαλιλαίου για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεν θα ήθελα να υπογραμμίσουμε τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του γιατί ζούμε σε έναν αλληλένδετο κόσμο και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διεθνή συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα συστήματα ραδιοπλοήγησης και για να μην έχουμε ανταγωνισμό στο διάστημα και γι' αυτό έχω υποβάλει τις τροπολογίες 13 και 14. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο τελευταίο κώδικα δεοντολογίας για τις δραστηριότητες ε, διαστήματος από τη Λέβη Άστον, αλλά δεν βρήκα τον κατάλληλο τρόπο να το κάνω. Γι' αυτό, αν συμφωνεί ο εισηγητής, μπορούμε να το κάνουμε με μια προφορική τροπολογία ή να ενταχθεί στο συμβιβασμό στους συμβασμούς 41 ή 42 της κυρίας Κρόνμπερκ. Όπως είπε και η κυρία Νικολάη στην τροπολογία 17, θεωρώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την ασφάλεια του συστήματος και στη 18 μιλώ για την ανάπτυξη δυνατοτήτων σε επίπεδο ΚΕΠΑ, έτσι ώστε να μην υποστούμε επιθέσεις στο ε, σήμα PRS. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης και με την τροπολογία 23 θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη διτή φύση του συστήματος. Επειδή υπάρχουν και συναφείς επιπτώσεις, θα πρέπει να δούμε να μας απασχολήσουν συστήματα διακυβέρνησης και λειτουργίας των συστημάτων, έτσι ώστε να βρίσκονται υπό πολιτικό έλεγχο και δεύτερον να τονίσουμε την ανάγκη για έλεγχο εξαγωγών. Βλέπω ότι στο τελευταίο θέμα συμφωνούμε με την κυρία Κρόμπερκ και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη δράση 2004-552 έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ μακριά και να δημιουργήσουμε την ε, εντύπωση ότι θέλουμε να επιβάλλουμε κανόνες στο Συμβούλιο. Τι εννοεί η κυρία Κρόμπερκ με την ε, τροπολογία 38. Πρόκειται για απόφαση του Συμβουλίου και ίσως ε, θα βρούμε άλλους τρόπους για να μιλήσουμε για τις προτιμήσεις μας μέσω επιστολής προς την ύπατη εκπρόσωπο ή να οργανώσουμε και μία ακρόαση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τις τροπολογίες που προβάλλουν άλλοι έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η κυρία Κρόμπεργκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν ως προς την 29 όπου μιλάμε για την απαλήφη του Union Security and Export Control, το ζητάμε όχι ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά θεωρούμε ότι δεν ε, έχει θέση εδώ. Θα θέλαμε μια τροπολογία που να ασχολείται με τον ε, κώδικα δεοντολογίας ως προς εξαγωγές όπλων και κανονισμούς διπλής χρήσης όταν διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να προτείνουμε μια ξεχωριστή τροπολογία. Άκουσα τα σχόλια σχόλια για την τροπολογία 38 που προτείναμε για την δράση 2004 κάθετος 552. Δεν θέλαμε εμείς να επιβάλλουμε αποφάσεις, αλλά να δούμε ότι σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης θα υπάρχει μία διαδικασία η οποία θα προβληθεί και θα επιβληθεί. Και θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να δώσουμε φωνή στις προτιμήσεις μας. Θα πρέπει να δούμε και θέματα διαστήματος, και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ασχοληθούν με το κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα και να δούμε κατά πόσο μπορεί να ανανεωθεί η συνθήκη για το διάστημα που χρονολογείται από το 67. Εδώ μιλάμε για ασφάλεια και ούτω καθεξής. Μιλάμε για ασφάλεια και άμυνα η οποία θα βρεθεί, θα αναπτυχθεί και στο διάστημα. Από πλευράς Κομισιόν θα ήθελε κάποιος να παρέμβει. Ευχαριστώ κύριε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να κάνω μια γενική παρατήρηση σε σχέση με μερικές τροπολογίες που προτείνονται για τη διτή χρήση ε, είναι ενδιαφέρον να μιλάει κανείς για δίτη χρήση στον κανονισμό, αλλά πιστεύουμε ότι ίσως θα έπρεπε να μην τονίσουμε τόσο πολύ αυτήν την πτυχή των πραγμάτων, δεδομένου ότι ούτως ή άλλως έχει ληφθεί μια απόφαση για τους όρους ε, πρόσβασης ε, στο σύστημα. δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Επίσης, σε κάποιες από τις τροπολογίες αναφέρεται να γίνεται αναφορά σε άλλα προγράμματα ή άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα στην 31 αναφέρεται το πρόγραμμα ε, Space Situational Awareness ε, ή αναφερόμαστε στην, στον κώδικα συμπεριφοράς. Πιστεύουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε σε αυτόν τον κανονισμό για αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες ε, ούτως ή άλλως είναι αντικείμενο άλλης νομοθεσίας. Τροπολογία 32. Σε αυτήν την τροπολογία πιστεύουμε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με την Κομισιόν και την ΙΕΣ e e γιατί η πρόταση είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποστήριξη ε, του, της ε, ε εξωτερικής υπηρεσίας, ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και όχι το αντίστροφο. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία 38 σε σχέση με την κοινή δράση, εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό το, το, το σύνολο του κειμένου για την κοινή δράση να αναφέρεται στη συγκεκριμένη τροπολογία και πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κυρία Άστον ε, έλαβε γνώση και ε, γνωστοποίησε στον κύριο Ταγιάννη ότι έχει σκοπό να ενημερώσει αυτήν την κοινή δράση δύο τεχνικές μάλλον λεπτομέρειες αλλά σημαντικές. Στην τροπολογία 18 αναφέρεται το spoofing του συστήματος. Το σύστημα όμως είναι ήδη ούτως ή άλλως ε, στεγανό σε αυτό το spoofing. Ε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι το spoofing θα έπρεπε να αντικατασταθεί με το jamming. Και στην τροπολογία 26 που μιλάει για τη διαχείριση των κρίσεων, τα κράτη-μέλη πρέπει να γνωρίζουμε ότι θέλουν ε, να έχουν την ε, πλήρη διαχείριση των ε, θεμάτων αυτών και δεν θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο αποφάσεις για το θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη θα διαχειριστούν αυτές τις περιπτώσεις κρίσεων. Αυτά ευχαριστώ. Αυτά είναι τα σχόλια για τις τροπολογίες των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως στην τροπολογία 28 και 38 που έχουν να κάνουν ε, με την ε, κατάσταση της κοινή δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υπηρεσία μας ε, έχουν επαφές εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, να επικαιροποιηθεί το κείμενο λόγω διαφόρων λόγων που έχουν αναφερθεί ήδη και επίση ε, πρέπει να σα πω ότι υπήρξε και ανταλλαγή επιστολών μεταξύ ε, του Αντιπροέδρου Ταγιάννη και τη ΥΠΑ ε, τη εκπροσώπου ότι η αναθεώρηση της κοινή δράσης πρέπει τώρα να λάβει χώρα. Έχουν ήδη λάβει χώρα συζητήσεις μεταξύ της υπηρεσίας μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε ένα πρώτο αποτέλεσμα στο σχετικά εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Η κυρία ε, Κρόμπακη θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Με ναι, ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω για την τροπολογία 32. Έχετε δίκιο, είναι ανάποδα, ανα, ανάποδα αναφέρονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνεπικουρούμενη από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης κλπ. Και, και αυτό αντίστροφο. Επίσης, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρεται και η εξωτερική ε, ε, πολιτική, γιατί είναι πολύ σημαντική η διάσταση αυτή τη εξωτερικής πολιτικής για τα θέματα αυτά. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Θέλουν άλλοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Κύριε Τερόμ, πώς θέλετε να συνοψίσετε. Νομίζω ότι υπάρχει κοινό έδαφος και σίγουρα μπορούμε να βρούμε κάποια λύση με τη βάση των παρατηρήσεων που άκουσα. Το βασικό ζήτημα θα είναι πόσο πολύ θα τονίσουμε τη διτή χρήση. Και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και θα συνεχίσουμε βέβαια και τους συμβιβασμούς όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις σας που είναι πολύ καλή αφετηρία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία της γνωμοδότησης αυτής ε, θα γίνει στο Στρασβούργο, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, στις 5 Ιουλίου. Η ΙΤΡΕ θα ψηφίσει για την έκθεση αυτή στις 6 Σεπτεμβρίου και η συζήτηση στην Ολομέλεια θα γίνει τον Οκτώβριο. Λοιπόν, ψάχνουμε τον κύριο Κυρίλοφ, γιατί είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης Για την εφαρμογή της νομοθεσίας του ενιαίου ουρανού, επί της ουσίας υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Μεταφορών. Αύριο θα το ψηφίσουμε αυτό το θέμα. Στις 9.30, εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Σας το λέω γιατί πρέπει να έχουμε απαρτία για να, μπορέσουμε να ψηφίσουμε αύριο το πρωί αυτό το κείμενο και βασίζομαι στην παρουσία σας. Έρχεται σε δύο λεπτά ο εισηγητής μας. Bien, Monsieur Kirillov, notre euh, rapporteur pour l'avis sur la mise en œuvre. Περνάμε λοιπόν ε, στη γνωμοδότηση για την εφαρμογή της νομοθεσίας του ενιαίου ουρανού. Κύριε Κυρίλοφ, έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. I'm sorry I had... Ευχαριστώ, συγγνώμη, έπρεπε να φύγω. είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί είχαμε και την ε, αντιπροσωπεία της, ε, του Αζερβαϊτζάν ε, και έπρεπε να τα συμβιβάσω όλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία. Θα ήθελα όλους να σας ευχαριστήσω, όλους όσους συμμετείχατε. Ειδικότερα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν κάποιες πολύ καλές τροπολογίες για τη γνωμοδότησή μου. 12 τροπολογίε μόνο λάβαμε, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει ιδιαίτερη συνένεση μεταξύ των Ευρωβουλευτών ε, και αυτό δείχνει ότι η Υποεπιτροπή κατανοεί τη σημασία της ε, στρατιωτικής ε, σημασίας του ενιαίου νερού και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας σύντομα. Η ασφαλής και ευέλικτη χρήση του ενιαίου ουρανού είναι δυνατή μόνο αν υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ ε, πολιτών και ε, ε, στρατιωτικών και πρέπει να βοηθηθεί, να διευκολυθεί η προσπάθεια αυτή όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρέπει το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται τακτικά ε, πώς εξελίσσεται η εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτός είναι ρόλο και της υποεπιτροπής μας και βεβαίως της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Η πρόκληση θα παραμείνει μετά την έγκριση της γνωμοδότησης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, η συγγήτρια, η κυρία Φώστερ, θα συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις απόψεις μας στην έκθεσή της. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους συναδέλφους να συζητήσουν με τους ε, ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Μεταφορών το θέμα αυτό για να εξασφαλίσουν ότι η γνωμοδότηση θα τύχει ευρεία αποδοχής γιατί αν τα στοιχεία που μας απασχολούν όλοι εμά δεν ληφθούν υπόψη σοβαρά, ε, θα υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για τη συνεισφορά και τη βοήθειά τη. Ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και την Eurocontrol. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει κύριε Πρόεδρε ότι, ένα, ότι, ότι ένας από τους βασικούς χρήστες ε, είναι... Ε, οι στρατιωτικές, ε, ο στρατιωτικός τομέας ε, και παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχε σε όλα τα επίπεδα των συζητήσεων και γι' αυτό άλλωστε πηγαίνει τόσο συχνά, τόσο αργά αυτή η διαδικασία, πρέπει να δούμε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά μας, γιατί η συνεισφορά μας Βεβαίως συμμετείχαμε στην όλη διαδικασία του ενιαίου ουρανού, όμως πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κάνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κυρίλοφ. Δεν βλέπω ιδιαίτερο πρόβλημα με τις τροπολογίες. Ένα ερώτημα όμως θα ήθελα να σας θέσω για την τροπολογία 8. Για ποιο λόγο θέλετε να διαγράψετε την αναφορά ε, στα αναμενόμενα ε, στρατιωτικά ε, έξοδα και θα ήθελα να ρωτήσω για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχετε καμιά πληροφορία κατά πόσο οι αεροπορικές δυνάμεις Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αναλάβουν το κόστος της συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ουρανό. Γιατί όπως αναφέρεται, το κείμενο, όπως αναφέρεται στο κείμενο γίνεται αναφορά στους στο κόστος και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να παραμείνει η αναφορά αυτή στο κόστος. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τις δαπάνες, η βιομηχανία πολιτικής αεροπορίας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτό το θέμα και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι επενδύσεις θα ανταποκριθούν ως προς το στρατιωτικό σκέλος. Το θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο τα αριθμητικά αυτά στοιχεία δεν είναι ακριβή. Αλλά κατανοούμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέλη της Ένωσης που χρησιμοποιούν στρατιωτικά αεροσκάφη εκτός Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση, να την ακολουθήσουμε για να βοηθήσουμε και τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε να απογειωθούμε ως προς τις δυνατότητες μας. Ο στρατηγός Λιλό έχει το λόγο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνας. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας ε, παρουσιάσω το ρόλο μας στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΖΑΡ. Θα ήθελα να αρχίσω υπογραμμίζοντας το ρόλο μας και να σας μιλήσω για το ε, αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στα κράτη-μέλη και να σας δώσω και ορισμένες υποδείξεις για το μέλλον. Θα ήθελα να πω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας έγκυται στο να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στη φάση εφαρμογής του προγράμματος ΣΕΖΑΡ. Στόχος είναι να μειώσουμε τις οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις στην αεροναυπηγική και να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες εφαρμογής του προγράμματος ε, ΣΕΖΑΡ. Αυτή η αποστολή βασίζεται σε τρεις ε, δράσεις. Η πρώτη αφορά τη σημασία, την αναγνώση της διάστασης του προβλήματος σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, ξεκινώντας από τους υπουργούς, από το Γενικό Στρατηγείο και α, κινούμενοι προς όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Θέλουμε να εναρμονίσουμε τις θέσεις μας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας άμυνας έτσι ώστε να μειωθούν ε, οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι και ως προς το πρόγραμμα αυτό που καμιά φορά απορρέουν. Η τρίτη αφορά τη διασφάλιση της συνεισφοράς της άμυνας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για την προετοιμασία της φάσης deployment. θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στην ε, εξάλληψη επικαλύψεων, στη συμπληρωματικότητα και στην αξιολόγηση της πείρας μας μέσα στα πλαίσια του UMS, UMC, Eurocontrol και NATO. Ως προς τις επιπτώσεις αυτής της δράσης, θα ήθελα να πω ότι με βάση αυτή τη δράση και χάρη σε εκείνη, η κοινότητα άμυνας είναι πιο καλά πληροφορημένη και εμπλεκόμενη και αυτό αφορά τα στρατηγία άμυνας των κρατών μελών που λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις του ΣΕΖΑΡ ως προς την ε, επιχρησιακή του δραστηριότητα. Και μία άλλη επίπτωση έχει σχέση με τη διασφάλιση τη συμμετοχής της άμυνας στα πλαίσια του deployment με βάση την ενδιάμεση επιτροπή deployment, η οποία ήδη συμμετέχει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετέχει και το στρατιωτικό σκέλος στην δραστηριότητα αυτή ανάπτυξης για να ορίσουμε και τον ε, στρατιωτικό συντονιστή ταχείας ανάπτυξης, της δύναμης ανάπτυξης, για να ορίσουμε κοινά σχέδια στρατιωτικού σκοπού και για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις οικονομικές δυνατότητες. Τέλος, μας ενδιαφέρει η υποστήριξη και ο ορισμός των ε, οικονομικών κινδύνων στο πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ και στα ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για, ε, ερω... για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Μήπως η Επιτροπή θέλει το λόγο. Όχι. Η κυρία Γκόμες. Κυρία Γκόμες, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμώ το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να δώσει μία όθηση στη συγκρότηση αυτού του συστήματος ΣΕΖΑΡ, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως προς την ασφάλεια του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Και πιστεύω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ε, έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο κεφαλαιόδου σημασίας στη συγκρότηση αυτού του συστήματος για να φτάσουμε και σε μία ανάλυση, μακροχρόνια ανάλυση, κάνοντας μία προβολή στο μέλλον σε σχέση με τις απειλές ε, στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Νομίζω ότι ο οργανισμός έχει λόγο ύπαρξης και θα πρέπει να υποστηρίξει το πρόγραμμα και τη λειτουργία του. Θα ήθελα να ρωτήσω τον στρατηγό ποιες θα είναι οι συνέπειες ή σε τι συμπεράσματα μπορούμε να φτάσουμε με βάση τα δεδομένα του 2007 όταν ε, έγιναν οι έρευνες για τις ε, πτήσεις της CIA που κατέδειξαν ότι υπήρχε μεγάλη αδυναμία ελέγχου του εναερίου μας χώρου και ως προς τους ελέγχους και ως προς την ασφάλεια. Όσον αφορά τις ε, πτήσεις του πολιτικού σκέλους, μπορούν κάτι να καταδείξουν ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, γιατί πρόσφατα μεταβήκαμε στη Λιθουανία μετά από τη διενέργεια αυτής της έρευνας και η Λιθουανία τότε δεν ήταν ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είχε λόγο να ακολουθήσει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλώντας όμως με τον ε, Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, είδαμε ότι αυτό που δεν υπήρχε στη Λιθουανία δεν υπήρχε ούτε καν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν είμαι σίγουρη ούτε καν ε, εάν στην Πορτογαλία που είναι κράτος μέλος εδώ και χρόνια, εάν υπάρχει αυτό το σκέλος. Μιλάμε για το PNR. Για τις ε, μη τακτικές πτήσεις δεν έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Μπορεί κανείς να μεταφέρει ό,τι θέλει, παιδιά, οτιδήποτε κανένας δεν ελέγχει και δεν υπάρχουν ε, ούτε καν κατάλογοι επιβατών και φροντίστων. Αυτό είναι απαράδεκτο, ασύλληπτο. Γιατί αν ε, ε, μπορούν να γίνουν μεταφορές ανθρώπων που θα βασανιστούν αλλού, τότε μπορεί να μεταφορθούν, να μεταφορθούν και ναρκωτικά και ούτω καθεξής. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον στρατηγό κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν ε, μέτρα ρύθμισης και στην πολιτική αεροπορία. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών αποκλειστικά. Θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση είναι πολύ καλή. Με τις νέες εξελίξεις που έχουμε τώρα, όπως τα drones, τα μη επανδρομένα αεροχήματα για τις επιλεκτικές θανατώσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο και ίσως κάποια μέρα θα μας πλήξουν και εμάς. Πρόσφατα, στον διάλογο με τους Αμερικανούς φίλους, Υπέβαλα αυτή την ερώτηση και μου είπαν ε, ότι υπό έκτακτες συνθήκες όλα επιτρέπονται. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μιλώ για χώρες, αλλά για ομάδες συμφερόντων που μπορούν να αγοράσουν drones και να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν υπερπτήσεις εκεί που θέλουν, πάνω από μια πρεσβεία, την Αμερικανική πρεσβεία, μια Αμερικανική πρεσβεία, μια Βρετανική στην Ευρώπη ή αλλού. Δεν ξέρω κατά πόσον κάτι τέτοιο θα αποτιμηθεί στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης ασφάλειας και μέσα στα πλαίσια του Σέζαρ και της εύρυθμης λειτουργίας του. Ο κύριος Λίζεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, διότι ούτως ή άλλως πολλά έχουν ήδη ηλεχθεί και εξ ονόματος του ΕΛΚΑ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κυριλόφ, διότι πραγματικά μπορέσαμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά ε, είμαστε γείτονες στις ε, Βρυξέλλες ε, και μετακινούμεθα με το ίδιο αυτοκίνητο. Άρα μπορούσαμε να συζητάμε και εντός και εκτός κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι, παρατηρήσεις της Επιτροπής μου θα γίνουν, ε, θα, θα, θα εισακουστούν και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία θα πρέπει να ακουστούν. Παραδείγματος χάρη στο σημείο 2 Λέμε ότι η χρησιμοποίηση του εναερίου χώρου, η χρήση του, του αερίου χώρου δεν πρέπει να αφορά μόνο τις στρατιωτικές αρχές, αλλά και άλλες υπηρεσίες, π.χ. την ακτοφυλακή, την πυροσβεστική, τους, ε, τα τελωνία. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε με πολλούς οργανισμούς και θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην ε, Επιτροπή. Αυτό το οποίο αναφέρουμε στο σημείο 5, δηλαδή η απαραίτητη συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Και χαίρομαι γιατί η συνεργασία αυτή βελτιώνεται. Εάν βελτιωθεί όμως, λέγεται εδώ ότι αν βελτιωθεί ε, πρέπει να βελτιωθεί. Αλλά διερωτώ με στο παρελθόν που... ποιο ήταν το πρόβλημα και τώρα βελτιώνεται. Όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε αφορούν το θέμα της ημέρας, αλλά μήπως μπορούσατε να απαντήσετε στα δύο τελευταία σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω όμως θα πρέπει να αναφερθώ στο... στην εντολή που έχει πάρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα καθήκοντα τα οποία ανέλαβε αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τους κανόνες που έχουν αποφασιστεί για την πολιτική αεροπορία. Και αυτό γίνεται υπό την αρμοδιότητα της ΕΑΣΑ. Εμείς λέμε ότι ο κανόνας ο τομέας μάλλον, ο στρατιωτικός που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτές ε, τις, αρμοδιο... τις ε, υποχρεώσεις αν θέλετε, θα πρέπει να σεβαστούν κάποιους κανόνες. Οι στρατιωτικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτούς ε, τους, αυτό το χώρο όπως σας είπα πρέπει να σεβαστούν αυτούς τους κανόνες και αυτή την, αυτά τα καθήκοντα τα οποία έχουμε, μας έχουν ανατεθεί. Τώρα για τα, τα drones, ε, η συμμετοχή μας περιορίζεται στον τεχνολογικό τομέα. Δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στα πλαίσια των κανόνων για την διαχείριση της πολιτικής αεροπορίας εάν αύριο υπάρξει μια εμπορική ανάγκη να ενταχθούν αυτά τα drones στην πολιτική αεροπορία τότε θα πρέπει να γίνει με βάση τις ε, τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες. Εκεί σταματάει η δική μας ε, αρμοδιότητα και τα δικά μας καθήκοντα. Δηλαδή εμείς πρέπει να σεβαστούμε απόλυτα τις εντολές που μας έχουν δώσει οι Υπουργοί μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΣΑΡ. Η Κομισιό μήπως θα ήθελε να θίξει το σημείο αυτό. Ευχαριστώ, δεν μπορώ να συνεχίσω στα Ιταλικά, διότι με τον τρόπο αυτό τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον στρατηγό, διότι με πρόλαβε και απήντησε και είπε πολλά από τα πράγματα τα οποία θα προσπαθήσω και εγώ να πω σύντομα. Καταρχάς είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την ασφάλεια. Όπως ε, και στην ε, προηγούμενη παρέμβαση που είχαμε κάνει εδώ στο Κοινοβούλιο για το ίδιο θέμα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην ασφάλεια του safety δηλαδή και του security. Αυτές οι δύο, όροι, safety και security, και που αφορούν ε, θέματα τελείως ε, διαφορετικά. Το, ο Ευρωπαϊκός Ενιαίος Ουρανός έχει να κάνει με θέματα ασφάλειας ε, όσον αφορά την, διαχείριση των, την ασφαλή διαχείριση των πτήσεων και των πολιτικών πτήσεων και των στρατιωτικών, διότι χρησιμοποιούμε τον ίδιο αέριο χώρο. Άρα θα μπορούσαμε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να κυκλοφορεί κανείς ασφαλώς σε αυτό το χώρο. Η βασική στόχοι του ενιαίου ευρωπαϊκού αγορα, ουρανού αφορά την αύξηση της ε, χωρητικότητας, ε, διότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, ε, μεγαλύτερη ανάγκη για αεροπορικές μεταφορές. Τώρα βέβαια λόγω της ύφεσης, οικονομικής ύφεσης, αυτή η αύξηση δεν είναι τόσο σημαντική όπως την προβλέπαμε στο παρελθόν και αφορά το, το επίπεδο, το συνολικό επίπεδο ασφάλειας και αυτό είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Αφορά επίσης ε, την, τις περιβαλλοντικές συνέπειες που έχουν οι αναέριες μεταφορές και έχει να κάνει επίσης ε, και με το, το θέμα της αποτελεσματικότητας κόστους. Όσον αφορά τώρα το θέμα της security, υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας που ε, αναθέτει το θέμα αυτό στο ΝΑΤΟ, κυρίως όσον αφορά την, ε, τις χώρες που αναγνωρίζει αυτή την ε, αρμοδιότητα. Και ο συνάδελφος στην τελευταία του ερώτηση αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε Δεν μπορούμε να μπούμε σε πολιτικές αναλύσεις αυτή τη στιγμή. Αυτή η συνεργασία όμως γίνεται σε τεχνικό επίπεδο. Και θα πρέπει να περιορίσουμε τον, ε, την, να περιορίσουμε τον αντίκτυπο στην διαλειτουργικότητα ε, των συστημάτων που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος τον οποίο ε, προσπαθούμε να υλοποιήσουμε και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας διότι προσπαθεί να ξεκινήσει να διευκολύνει αυτό τον διάλογο έτσι ώστε να είναι ε, δυνατό, δυνατή αυτή η συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο. Ε, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Τώρα για τα drones να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή ε, αυτές τις εβδομάδες ξεκινάει μία πρωτοβουλία που έχει σαν στόχο να διευκολύνει ένα συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να ενταχθούν αυτά τα συστήματα τα οποία έχουν πολιτικό στόχο κυρίως να ενταχθούν στον, ευρω... ευρωπαϊκό χώρο, στον ευρωπαϊκό ουρανό. Υπάρχουν ε, πολλές χρήσεις ε, ε, αυτών των drones και ελπίζουμε ότι θα υποφεληθεί η Ευρώπη από αυτές τις πολλαπλές χρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυριλόφο. Πρόεδρε, συμφωνώ. Και εγώ συμφωνώ. Εγώ ήμουν ικανοποιημένο όταν είδα στι αρχικέ διαβουλεύσει ότι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα παίζει ένα χρήσιμο ρόλο σε αυτό το συντονισμό. και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων η συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες από τον ΝΑΤΟ είναι χρήσιμη, επικοδομητική, παραγωγική και θα έπρεπε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά τέλος πάντων όταν γίνονται πολιτικά πια τα ζητήματα αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα. Τώρα, πώς θα χρησιμοποιηθεί η γνωμοδότησή μας ε, στην Επιτροπή Μεταφορών. Εγώ είχα μια καλή συζήτηση με την εισηγήτρια, την κυρία Φώστερ, εξέφρασε κάποιες αντιρρήσεις σε σχέση με το μακροσκελές κείμενο που προτείνουμε και χαίρομαι που οι συνάδελφοι με προσπάθησαν να το συντομεύσουν. Προσπαθώ να τονίσω το σημαντικό στοιχείο της στρατιωτικής πτυχής και ελπίζω, ελπίζω ότι κάποιες από τις προτάσεις μας, αρκετές από τις προτάσεις μας ε, θα ενσωματωθούν. Νομίζω ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους μας στην Επιτροπή εκείνη και να ζητήσουμε την υποστήριξή τους. Ελπίζω ότι το σημαντικότερο τμήμα της ονομοδότησής μας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Οπότε τελειώνει η συζήτηση ε, για αυτό το θέμα σήμερα. Αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε στις 9.30 επί της γνωμοδοτήσεως αυτής για έγκριση στη συνέχεια στην Επιτροπή Μεταφορών ε, που θα παρουσιαστεί στις 9 και 10 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μείνουμε εδώ για σήμερα. Ε, θα ήθελα να ζητήσω μόνο από τους συντονιστές των ομάδων να παραμείνουν. Ε, θα κάνουμε μια συνεδρίαση του προεδρίου και κλεισμένων των θυρών. Ευχαριστώ πολύ.